Okay, colleagues, Πάμε αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μαραθώνιες προσπάθειες τις οποίες θα πρέπει να καταβάλουμε. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από τους ε, συντονιστές και από τις γραμματείες των πολιτικών ομάδων να θυμίσουν σε όλο τον κόσμο να φέρουν τις κάρτες ε, ψηφοφορίας τους γιατί χωρίς ε, κάρτες ψηφοφορίας δεν μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορίες. Μπορούμε να εγκρίνουμε τώρα την ημερήσια διάταξη που έχετε μπροστά σας. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις εντάξει. Έγκριση των πρακτικών 30 και 31 ε, Αυγούστου καθώς και 8 Σεπτεμβρίου. Έχετε κάποιες αντιρρήσεις ερωτήσεις. Αλλιώς τα εγκρίνουμε και αυτά. Και ερχόμαστε στον ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο, εξέταση τροπολογιών. Η κυρία Σερακιάνη είναι η, η Η Δέμπρα όταν είσαι έτοιμη, σου δίνω το λόγο όταν είσαι έτοιμη. Η κυρία Σερακιάνη, λοιπόν. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά ήταν μια πολύ δεσμευτική υποχρέωση. Έχουμε 18 συμβιβαστικά κείμενα και μια σειρά από τροπολογίες. Είδατε πόσο ε, παχυλός είναι ο κατάλογος ψηφοφορίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, για τη συνεργασία αυτούς τους μήνες. Πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό, πόσο μάλλον για ένα θέμα τόσο ε, σημαντικό και πολύπλοκο όπως το Recast. Να σας ε, θυμίσω μερικά σημαντικά σημεία για το σιδηροδρομικό Recast συμπεριλαμβάνει τα άρθρα 55 ως 57 που είναι πολύ ρυθμιστικά, είναι εντελώς ε, ε, δεσμευτικά. Εμείς προβλέψαμε τη δημιουργία ενός δικτύου εργαζομένων με την συμμετοχή της Κομισιόν για να τους βοηθήσει στις εργασίες και στις αποφάσεις προσπαθήσαμε να καταστήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατική. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Κομισιόν να ε, προχωρήσει στην, σε μία πρόταση για τον Ευρωπαίο ρυθμιστή πριν από το 2014. Τώρα για τα άρθρα 13 παράρτημα 3 σχετικά με τη σιδηροδρομική επαναδιατύπωση εμείς ε, για την παροχή ζητάμε αυτονομία των ε, σιδηροδρομικών οργανισμών όχι νομικά αλλά αποφασιστικά και νομικά. Ζητήσαμε επίσης ε, αυτονομία για το νίκιο και το leasing εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται για ένα χρόνο σχετικά με τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών υποδομών ε, και των ρυθμιστή ε, τονίσαμε ότι χρειάζεται ενίσχυση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη χρηματοδότηση των υποδομών και τα χρόνια, τα χρόνια που συνδέονται στην αναπτυξιακή στρατηγική είναι πλέον 7, η Κομισιόν πρόβλεπε 5. Όπως επίσης εισάγαμε και την υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να καλύπτουν τα χρέη του διαχειριστή των υποδομών όταν τα έσοδα δεν ανταποκρίνονται στον, στη χρηματοδότηση των, των σχεδίων, των προγραμματισμένων σχεδίων. Επίσης βάλαμε κίνητρα για την μείωση του θορύβου. Δεν τη συνδέσαμε με, με την ε, οδηγία για το ευρωσήμα. Θελήσαμε να αποφύγουμε αρνητικές επιπτώσεις ε, οικονομικές επιπτώσεις στον διαχειριστή της υποδομής για να μην έχουμε ε, κακές επιπτώσεις στις επενδύσεις. Μιλήσαμε για τις απεργίες στο παράρτημα 7 και τις ελάχιστες υπηρεσίες. Ξαναβάλαμε το κοινωνικό κέρδος στο άμεσο κόστος των σιδηροδρομικών υπηρεσιών μειώσαμε τις εκπτώσεις για τα τρένα, για τα ITCS και δώσαμε επίσης ε, κατευθύνσεις ε, για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε άλλα τμήματα της αγοράς. Επίσης, ε, θελήσαμε να προχωρήσουμε σε σχεδιασμό ικανοτήτων και δυνατοτήτων μόνο για τις βαλτικές χώρες. Τώρα στο άρθρο 15 προβλέψαμε να εμπλακούν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σίδηροδρόμων στον ελεγκτικό τομέα της Κομισιόν. Και γι' αυτό για να μπορέσουν να ελέγξουν το άνοιγμα τη αγορά στι σιδηροδρομικέ υπηρεσίε. Μετά έχουμε το άρθρο 6 για το διαχωρισμό των λογαριασμών που είναι ε, καρπό συμβιβαστικού κειμένου όπου εμεί ενισχύσαμε τον διαχωρισμό των λογαριασμών αποφεύγοντας τις ε, χρηματοπιστωτικέ μεταφορέ από τις υποδομές την λειτουργικότητα τη υπηρεσία. Πρέπει να σα πω ότι γι' αυτό το άρθρο Υπάρχει ένα, τμήμα το οποίο μας ζητήθηκε από το ΕΛΚ με το οποίο εγώ δεν συμφωνώ με το τελευταίο τμήμα του άρθρου 6. Υποστηρίζω ότι εμείς εργαστήκαμε για να μπορέσουμε να καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο διαφανή τον διαχωρισμό των λογαριασμών και εδώ θέτουμε όρους για να προχωρήσουμε στον χωρισμό των λογαριασμών. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει το αρχικό συμβιβαστικό κείμενο χωρίς ε, αυτήν την τροποποίηση. Εγώ θα καταψηφίσω λοιπόν αυτήν την τροπολογία. Για το άρθρο 7 και εδώ έχουμε ένα συμβιβαστικό κείμενο. Εμείς προσπαθήσαμε να τακτοποιήσουμε την ισότιμη πρόσβαση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, ανεξαρτησία σε νομικό επίπεδο οργανωτικό και αποφασιστικό του διαχειριστή της υποδομή, των υποδομών και ζητήσαμε από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει μία πρόταση μέχρι τις 31 2012 σχετικά με τον διαχωρισμό μεταξύ του διαχειριστή της υποδομής και του ε, διαχειριστή της υπηρεσίας. Εμείς ε, θέλουμε να μειώσουμε τις ε, τις εξουσιοδοτήσεις. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν από την Κομισιόν να μας πει τη γνώμη της για την τροπολογία 357 στο άρθρο 9 που παρουσίασε η κυρία Τικάου διότι έχω μερικές αμφιβολίες για αυτό το σημείο και θα ήθελα να ακούσω τις εξηγήσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τη Γραμματεία, πιο συγκεκριμένα τον Γιούργεν και τον Νταβίντ για τη δουλειά τους. very much, Ευχαριστώ πολύ κυρία Σερικιάνη. Ο κύριος Κούν για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Σερακιάνη, την εισηγήτρια. Ήταν Ηράκλειο το έργο της με την πραγματική έννοια της λέξης για να μπορέσει να επιτύχει οι συμβαστικές λύσεις μεταξύ μας. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε πραγματικά νέες κινήσεις σε σχέση με τους σιδηροδρόμους, φιλελευθεροποίηση γενικά, αλλά και παρόμοιες προδιαγραφές για όλες τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει υπό την αιγίδα ενός κοινού ρυθμιστικού σώματος. Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι χρηματικές, ε, ε, χρηματοδοτικές δυνατότητες των σιδηροδρόμων είναι κάτι το οποίο μπορεί τώρα να ελέγχεται και να αποτελεί αντικείμενο ταχαίων αποφάσεων από τι ρυθμιστικέ αρχές, ώστε να μπορέσει να υπάρξει η σωστή συμμετοχή των συνδοτομικών εταιριών σε όλες αυτές τις καινοτομίε. Πρέπει ακόμα να ληφθούν οι αποφάσεις για τις ουσιαστικές υπηρεσίες, τις ε, ελάχιστες υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, πόσο συχνά θα πρέπει να έχει ο καθένας τέτοιες βασικές υπηρεσίες σιδηροδρομικές, σε ποιο βαθμό αυτό πρέπει να είναι ένα τμήμα των υποχρεώσεων κάθε σιδηροδρομικής εταιρεία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι θετικό να υποχρεώσει κανείς αμέσως μια εταιρεία να ακολουθήσει το σύνθημα use it or lose it, δηλαδή άμα δεν χρησιμοποιεί μια σιδηροδρομική γραμμή να πρέπει να την πουλήσει, να τη δώσει σε κάποιον άλλο. Κάτι άλλο το οποίο είναι απαραίτητο για μένα για να εξασφαλίσουμε ένα θεμητό ανταγωνισμό είναι ο τρόπος καθορισμού των τιμολογίων και των ε, κομίστρων. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τι, ποια είναι τα, ποιες είναι οι συνιστώσεις αυτών των ε, τιμών και του κόστους μιας συνδρομικής επιχείρησης, γιατί μόνο σε αυτό μπορεί να βασιστεί ο ανταγωνισμός. Και νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε όλοι μία συνένεση στο θέμα αυτό, ώστε πρέπει να υπάρξει μια χωριστή λογιστική μεταξύ της διαχείρισης των υποδομών και της λειτουργικής ε, πλευράς μιας ε, επιχειρήσης. Να υπάρχει μια σαφής διάκριση λοιπόν, και εδώ έρχομαι στο άρθρο 6 παράγραφος 4, Φυσικά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι και για την χρηματοδότηση των υποδομών είναι απαραίτητες πιστώσεις από μια εταιρεία η οποία έχει την διαχείριση ε, των γραμμών ή από κάποιους επενδυτές οι οποίοι συμμετέχουν και κάποιος πρέπει να αποσβέσει το κόστος αυτών των επενδύσεων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο για μας το άρθρο 6 παράγραφος 4 το αντιμετωπίσαμε με αυτή την οπτική γωνία. Αλλά είναι σημαντικό επίσης να θελήσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα διαμιάς όπως λέμε και στις αιτιολογικές ε, σκέψεις θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Κομισιόν η Κομισιόν θέλει να ξεκινήσει με μία πρόταση την ε, ιδέα αυτή του διαχωρισμού του διαχειριστή των υποδομών από την εταιρεία. Να ξεκινήσει λοιπόν η προβληματική και η διαβούλευση για τα θέματα αυτά τον επόμενο χρόνο και να συνεχίσει πάντα με το στόχο ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα εμπορεύματα, όσο το δυνατόν περισσότεροι επιβάτες θα μπουν σε σιδηροτροχές ως τρόπος του λέγει και ως πραγματικότητα και αυτό θα προωθήσει μια πιο οικολογική μορφή μεταφοράς και θα μπορέσει να επιτρέψει και στα εμπορεύματα και στους ανθρώπους να φτάνουν στον προορισμό τους. Ευχαριστώ. Τρεμόσο. Ευχαριστούμε αν μπορείτε να είστε σύντομος. Πρόεδρε, από τη συνάδελφη, τα καταφέραμε τελικώς με ένα πολύ τεχνικό φάκελο. Συγχαρητήρια καταρχήν στην εισηγητρία, διότι δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί συμβασμός. Η ζωή της δεν ήταν εύκολη, όπως λέμε, παρά τις εντάσεις και την ασυνοησία μετά από σειρά συσκέψεων, καταλήξαμε σε συμβασμό σε σειρά θεμάτων. Κατανοώ τις της Προεδρίας και της Γραμματείας για την ψηφορία αύριο. Ζήτησαμε όμως ξεχωριστές ε, ψηφορίες για το 13 και το 7 για τις συμβαστικές ψηφορίες. Στην τελική λίστα αυτά έγιναν προφορικές τροπολογίες. Δεν ξέρω αν θέλετε να αλλάξετε κάτι. Εάν δεν καταστεί δηλαδή η ξεχωριστή ψηφορία, τώρα θα ζητήσουμε ξεχωριστή ψηφορία για ολόκληρη την παράγραφο. Από τη συνάδελφη να πω επίση ότι οι φιλελεύθεροι ανέκαθεν διαπραγματεύονται επικοδομητικά για να διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνία. Σε πολλέ περιπτώσει οι φιλελεύθεροι πιστεύω ότι συνέβαλαν προ τούτο. Και τούτο διότι η στάση μα ήταν αυτό συνεπή. Από την αρχή, από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Θα έλεγα μάλιστα μέχρι και σήμερα. Από την πρώτη συζήτηση, οι προτεραιότητε των φιλελευθέρων ήταν η απελευθέρωση της αγοράς και η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή. Εμείς από μια περίκλειστη χώρα όπου το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών συγκρίνονται συνεχώς, για μας οι αρχές αυτές είναι ζωτική σημασίας. Να σταματήσουμε δηλαδή τον μπλοκάρισμα του ανταγωνισμού και τα εμπόδια στον ανταγωνισμό από χώρα σε χώρα. Προς τούτο χρειαζόμαστε ένα, μια ισχυρή ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Και τούτο επιτυγχάνεται με το 57α. Με τη δημιουργία δηλαδή μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή σε δύο χρόνια από τώρα. Από την άποψη αυτή εκφράζουμε την ικανοποίησή μα τι τροπολογίε για τα άρθρα 55-57, για τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ και τι αρμοδιότητέ του. Ενισχύεται έτσι οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ανεξάρτητη Αρχή και χαιρόμαστε βεβαίω το ότι οι χρεώσει είναι συνάρτηση των συνδικών της αγοράς. Στο 55, στο 55 χαίρομαι που προσθέθηκε κείμενο το οποίο λέει ότι ο πρόεδρος και οι αρχές της Εθνικής Εθνικής Αρχής θα ορίζονται από τα εθνικά κοινοβουλία. Για μένα και την κυρία Μπιλμπάου αυτό ήταν ένα σημείο ζωτικής σημασίας. Για το άνοιγμα τη αγορά, θέλαμε να περιλάβουμε στην αδιατύπωση, στο 7, στην παράγραφο 3, να υπενθυμίσουμε στην Κομισιόν να υποβάλει προτάσει ω το τέλο του 2012. Ως φιλελεύθερη επίσης ζητήσαμε ξεχωριστή ψηφοφορία για το τέλο τη πρόταση. ήμασταν και είμαστε κατά του παρακτήματος 8, γιατί για εμάς δεν είναι λογικό το άμεσο κόστος του τρένου να συμπεριλαμβάνει ε, τα σχολεία, τα εστιατόρια, τους παιδικούς σταθμούς και τις συντάξεις όλων των υπαλλήλων των σιδηροδρόμων. Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει τον τομέα, να γίνει δηλαδή πιο ανταγωνιστικός σε σχέση, ή σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς. Και εκπλησόμεθα ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει μια τέτοια πρόταση. Επίση, Θα θέλαμε την ελάχιστη, την βασική υπηρεσία να εξασφαλίζεται στην περίπτωση απεριών που είναι εις βάρος των καταναλωτών και της οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώς ζητούμε χωριστή ψηφορία για την παράγραφο 9 του παραρτήματος 7. Τέλος, όσον αφορά την αποδέσμευση και τη σχετική συζήτηση και επειδή δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε όλο το πακέτο, για το θέμα της αποδέσμευσης, επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ του να μείνει έξω από την αναδιατύπωση και αναμένω του χρόνου την πρόταση, τη σχετική πρόταση της Κομισιόν. Επίσης, δεν έχω κάπου καταλήξει ως προς αυτό, ούτε έχω ιδολική θέση. Θα ακούσω τα επιχειρήματα των άλλων πλευρών ενώπιση του μέλλοντος. Εάν δηλαδή το άνοιγμα της αγοράς, η επιτυχάνεται έτσι καλύτερα με ξεχωριστό τρόπο. Επίσης, το εκτιμώντας 11, έχουμε την τροπολογία 174. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την υποστήριξή της. Τέλος, στο άρθρο 6, 4, πρέπει να πω ότι ακόμη και αυτή την εβδομάδα είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ με την συμπερίληψη όμως της τελευταίας τροπολογίας, με την οποία όμως, αν δεν κάνω λάθος, είναι κατά η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Ζήλ, να σας δώσω μια εξήγηση όσον αφορά το έτοιμά σα. για τροπολογία επί της επισήμως αποδεκτής τροπολογίας. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε μια τροπολογία που είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού με γραπτή τροπολογία εκτός εάν έχετε τη σύμφωνη γνώμη όλων όσων έχουν επιτύχει τον συμβιβασμό. Μπορείτε να θέλετε να την παρουσιάσετε ξεχωριστά ή να την υποβάλλετε ως προφορική τροπολογία. Αλλά δεν μπορείτε να υποβάλλετε, επαναλαμβάνω, γραπτό επίσημη τροπολογία για κάτι, για μια τροπολογία, η οποία είναι αποτέλεσμα συμβασμού. Γι' αυτό το λόγο κρίναμε ότι βάσει του 163, του κανόνα 163, δεν μπορείτε να υποβάλλετε την τροπολογία όπως περιέγραψα. Οπότε, το έτοιμά σα περί της προσθήκης τη λέξης legal θα πάρει τη μορφή προφορικής τροπολογία. Ελπίζω να μην έχει κανεί αντίρρηση. Επ' αυτή θα ψηφίσουμε τη προφορική επειδή, επαναλαμβάνω, έγινε ότι έγινε χωρί την σύμφωνη γνώμη των ομάδων που είχαν καταλήξει σε συμβασμό. Αυτή είναι η εξήγηση για την οποία ε, κάνω την τροπολογία σας ως προφορική. Τώρα να προετοιμάσω τον κατάλογο τροπολογιών μην νομίζετε είναι εύκολο. και Ζηλέα, από την ECR. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές. Ξέρουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε δυσκολίες είχαμε πολλά προβλήματα το καλοκαίρι, τώρα το φθινόπωρο έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και έχουμε καταφέρει να φτάσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό συμβαστικών τροπολογιών από ό,τι φανταζόμασταν το καλοκαίρι. Για πολλές από αυτές τις συμβαστικές λύσεις θα τις υποστηρίξουμε στην ομάδα των συντηρητικών, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, παρά το γεγονός ότι ορισμένες από τις τροπολογίες μας εμείς θεωρούμε ότι είναι πιο εύστοχες από αυτά που περιλαμβάνουν οι συμβαστικέ λύσεις. Θέλουμε η Κομισιόν να καταλήξει σε κάποιες προτάσεις μέχρι το τέλος του 2012 για την αποδεσμοποίηση. Εγώ συμφωνώ τώρα σε ορισμένα σημεία με αυτά που είπε ο συνάδελφός μου από το... τους φιλελεύθερους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη συμβαστική τροπολογία ε, γιατί σε περίπτωση απεριών πρέπει να διατηρείται η ελάχιστη υπηρεσία και επίσης τις τροπολογίες Q που αφορά τις ε, κοινωνικές παροχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ως τμήμα των άμεσων, <clears throat> του άμεσου κόστους μιας επιχείρησης. Κοινωνικές αυτές υπηρεσίες, και ηλικία κτλ. Όλα αυτά δεν πρέπει να καταλογίζονται ως άμεσο κόστος. Επίσης για τους εθνικούς ε, ρυθμιστές και την ε, δημιουργία δικτύων έχουμε ένα σχόλιο από την δική μου πολιτική ομάδα. Η Κομισιόν δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην διακυβέρνηση αυτών των υπηρεσίων διαδικτύωσης, δικτύωσης, αλλά θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάποιες συμβαστικές ιδέες εδώ. Αυτή είναι λοιπόν η θέση της ομάδας μας <clears throat> και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν υπόψη της ιδιαιτερότητας της αγοράς της Βαλτικής και την δυσκολία που μπορεί να υπάρξει στο να καθοριστεί το τίμημα για τους χρήστες των υποδομών. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. η πρόταση των πρασίνων δεν την έχω παρακολουθήσει πλήρως για, την, για το, την απόλυτο διαχωρισμό που χρειάζεται. για την ε, λειτουργία των σιδηροδρόμων οι οποίοι μπορεί να, έχουν, να διακινούν προς τρίτες χώρες αλλά εν θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Κράμερ να μας παρουσιάσει την άποψη των Πρασίνων για το θέμα αυτό. Αυτά λοιπόν από τη δική μου πλευρά και πάλι ευχαριστώ την Τέμπορα και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Κράμερ για τους ε, πράσινους. Και εσείς τέσσερα λεφτά παρακαλώ. Ναι. <clears throat> και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να καταλήξουμε στον ε, στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Η οδηγία της Κομισιόν δεν είχε καταρχήν τίποτα για την αποδεσμοποίηση δεν είχε τίποτα ε, για, το άνοιγμα της επιβατικής, των επιβατικών συνδρομικών γραμμών. Ήταν απλώς μια μικρή τροποποίηση του πρώτου πακέτου για τα συνδρομικά θέματα. Ξέρουμε στην Ευρώπη ότι υπάρχει πρόβλημα με πολλές αγορές οι οποίες είναι κλειστές, αλλά δεν εξαρτάται από το αν υπάρχει η απόλυτη διάκριση μεταξύ λειτουργικής δραστηριότητας και υποδομής που θα καθορίσει μια ε, επιχείρηση αν είναι κλειστή ή όχι. Στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη, υπάρχει αυτή η διάκριση, αλλά η αγορά είναι κλειστή στα Πυρηναία. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρέμβαση. Σε άλλε χώρε υπάρχει μια διάκριση η οποία δεν έχει προχωρήσει πλήρω, αλλά παρόλα αυτά η αγορά είναι ανοιχτή. Ο στόχο μα είναι πραγματικά να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την εθνικιστική στάση στους Ευρωπαίους, ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, να έχουμε μια ευρωπαϊκή πραγματικα να μπορεσουμε να ξεπερασουμε την εθνικιστικη σταση στου ευρωπαϊκού ευρωπαικους να εχουμε μια ευρωπαικη προσεγγιση και αυτό ξεκίνησε ήδη μόνο το 2007 με τις εμπορευματικές μεταφορές, θέλουμε να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις και η δυνατότητα ορισμένων εταιριών να κλείνουν την αγορά προς όφελός τους. Γι' αυτό θέλουμε ο, <clears throat> ο να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την ε, δυνατότητα πρόσβασης ή μη πρόσβασης σιδηροδρομικών εταιριών στην αγορά. Και αυτό πρέπει να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο, γιατί σε ορισμένε χώρε μπορεί να χρειαστεί να αποφασίσει ένα ρυθμιστή, αλλού κάνει δύο εβδομάδε, αλλού κάνει δύο χρόνια. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια σαφή διαδικασία, ώστε να ξέρει κανεί πραγματικά τι θα προκύψει. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μια ενιαία ρυθμιστική διαδικασία για το πλήρε άνοιγμα τη αγορά των σιδηροδρόμων. Και από την πλευρά τη Κομισιόν έχουμε την ε, απόφαση που εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην οποία πρέπει να απαντήσει η Κομισιόν και μετά από πολλές συζητήσεις νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η Κομισιόν μέχρι το τέλος του 2012 να δώσει κάποια πρόταση για την αποδεσμοποίηση και για το άνοιγμα των επιβατικών μεταφορών. Και είναι σημαντικό και στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια σαφής εστίαση Στι ρυθμιστικέ δραστηριότητε, δραστηριότητες, γιατί ήταν πολλά κράτη-μέλη που λένε βεβαίω να διαχωρίσουμε τι υποδομέ από τι μεταφορικέ δραστηριότητε, αλλά η ρύθμιση είναι θέμα το οποίο θα το αφήσετε σε εμά. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα και όχι η λειτουργική, η λειτουργική διαχωριστική αυτή η δράση. Για τον Ζήλε, εμεί πάντα σα υποστηρίζουμε γιατί ξέρουμε ποια είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα στη Βαλτική, αλλά υπάρχουν και περαιτέρω προβλήματα μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδος και Τουρκίας, γιατί εκεί παρεμβαίνει μια τρίτη χώρα και δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς εναλλακτικέ γραμμές. Πρέπει να χρησιμοποιήσει τις ίδιες γραμμές αυτές. Όταν τα πράγματα αφορούνται, αφορούν τρίτες χώρες, ε, υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση, αλλά πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα με το εύρος των γραμμών όταν υπάρχει μια τρίτη χώρα. Αυτό το οποίο εμεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι θα υπάρχει μια συμφωνία για το εύρος των γραμμών με άλλες χώρες ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε ότι έχουμε ακόμα προβλήματα μεταξύ Σερβίας, Βουλγαρίας, ε, Σερβία, με Βουλγαρίας, Ρουμανίας κτλ. Μπορούμε λοιπόν μέσα σε συμβαστικές λύσεις να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, ακόμα και δεν το έχουμε επιτύχει ακόμα. Λοιπόν, εν κατακλείδη, μπορώ να δεχτώ όλα αυτά. Αυτό το οποίο με ενοχλεί ακόμα είναι ότι, <clears throat> κύριε Μπάχ, δεν είναι για κοινωνικούς λόγους που το κόστος των ε, παιδικών σταθμών πρέπει να συμπεριληφθεί. Αλλά το απαραίτητο είναι όλες οι επιχειρήσεις να έχουν τις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού. Αν βάλουμε όλα αυτά τα κοινωνικά, το κοινωνικό κόστος στο τιμολόγιο για τους επιβάτες, τελικά δεν θα παίρνει κανείς το τρένο, θα παίρνει μόνο το αεροπλάνο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως. Αν συγκρίνουμε τα λεωφορεία με τα, με τα τρένα, οι εταιρείε λεωφορείων πρέπει να λάβουν υπόψη το κοινωνικό κόστος, αλλά δεν έχουν κόστος για την ε, στάθμευση των ε, οχημάτων τους και δεν έχουν τις ε, επιδοτήσεις και τις ελαφρύνσεις που έχουν τα λεωφορεία στη Γερμανία οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Αν λοιπόν τα λεωφορεία έχουν καλύτερη ανταγωνιστική θέση και από την άλλη πλευρά εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε το περιβάλλον, αυτό δεν βγάζει νόημα. Λοιπόν, ή όλοι πρέπει να πληρώνουν το κοινωνικό κόστος ή κανένα. Αλλά όχι οι σιδηρόδρομοι να πληρώνουν, να μεταφέρουν στον καταναλωτή το κοινωνικό κόστος και οι άλλε μορφέ μεταφορών όχι. Ευχαριστώ. Κόλτσα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εκπλήττομαι με τα όσα ακούω. Μήπως κάποιοι ήρθαν σε λάθος αίθουσα. Η δουλειά μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση των σιδηροδρόμων. Δεν είναι να αποδεσμεύσουμε να ξεχωρίσουμε πιβατική κίνηση, φορτία κλπ. Η βασική μας δουλειά είναι να βελτιώσουμε τη θέση των σιδηροδρόμων εν γέννη. Δυστυχώ η πρώτη δέσμη, το πρώτο πακέτο, δεν έχει διατυπωθεί σωστά και ανεβαίνει σε αυτόν τον σκοπό. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τους συναδέλφου. που λένε ότι η ίδια Κομισιόν πρέπει να θέσει προθεσμίες για την αποδέσμευση κλπ. Κοιτάξτε, όπου έγινε, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Ήταν καταστροφικά για τον σιδηρόδρομο, ο οποίος έγινε λιγότερο ανταγωνιστικός, ακριβώς διότι το κόστος ανέβηκε. Και είναι λογικό. Τρεις επιχειρήσεις στη θέση μιας έχουν ως αποτέλεσμα τριπλασιασμό του κόστους. Τώρα το αν το κοινωνικό κόστος πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη είναι θέμα συζήτησης. Ούτως ή άλλως τα στοιχεία του κόστους κάπου συμπεριλαμβάνονται. Αν έχετε πρόβλημα με αυτό, δεν πρέπει να τρώτε ούτε στις καντίνες, ούτε στα εστιατόρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση όπου έγιναν αυτά, μειώθηκε το μερίδιο των σιδηροδρόμων στις μεταφορές. Υποτίθεται κατά τα άλλα ότι το 2012 η Κομισιόν πρέπει να θεσπίσει τον πλήρη διαχωρισμό, την πλήρη αποδέσμευση. Αυτά τα μέτρα δεν έχουν θέση στο πακέτο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η οδηγία πρέπει να βελτιωθεί και όχι να απορριφθεί, να εξελιχθεί εντελώς αν θέλουμε να βελτιώσουμε την θέση των σιδηροδρόμων. Ας το σκεφτούμε λοιπόν καλύτερα. Χρειαζόμαστε βεβαίως ρυθμιστικές αρχές παντού σε όλους τους τομείς, αλλά δεν ξέρω αν έχετε πείρα από τους σιδηροδρόμους στη χώρα σας, αλλά οι υποδομές και η διαχείριση των υπηρεσιών πρέπει να είναι σε αρμονία. Αλλιώς θα γίνει αυτό το οποίο έγινε με τους αυτοκινοδρόμους, με τελείωτα μποτιλιαρίσματα, ιδιαίτερα σε ορισμένα σημεία, χωρίς σταθερές ε, ροές και σταθερές ταχύτητες στις οδικές μεταφορές. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Το ότι 20 χώρες δεν έχουν υλοποιήσει το πρώτο πακέτο, κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το πρώτο πακέτο. Οπότε, επαναλαμβάνω, επαληθεύστε τα δεδομένα και προσέξτε και δείτε τι έγινε εκεί που έγινε η αποδέσμευση. Δείτε τα καταστροφικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οκτώ ομιλητέ έχουμε ακόμη, συν την Κομισιόν, συν ε, την εισηγήτρια και μας μένουν μόνο 25 λεπτά. Επειδή δεν άκουσα καινούργια πράγματα, θα παρακαλέσω του επόμενου ομιλητές να τηρήσουν τον κανόνα των δύο λεπτών. Παρακαλώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια <clears throat> για την υπομονή που έδειξε στη συνεργασία μαζί της και για την διαθεσιμότητα να μπορέσει να ακούσει τις απόψεις όλων και να προχωρήσει εστιάζοντας την ανάγκη μιας καλύτερης και πιο έντονης ρύθμισης ώστε να εξοικονομήσουμε ενέργεια για τα άλλα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Έχουμε τώρα ένα τεράστια δύσκολο κατάλογο ψηφοφοριών, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πήρα πάλι πολλά ερωτήματα μέσα από την πολιτική μου ομάδα σε σχέση με τις πρόσθετες προφορικές τροποποιήσεις. Πιστεύουμε στο ΕΛΚ ότι μεταξύ την ε, τωρινή ψηφοφορία και την ε, Ολομέλεια μπορούμε να φέρουμε κάποιες ε, Αλλαγέ, αλλά δεν πρέπει να περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα και πιστεύω ότι πέραν από αυτέ που έχουν γίνει γνωστέ, δεν πρέπει να δεχτούμε καθόλου περαιτέρω προφορικέ ε, τροποποίησεις. Αυτή νομίζω ότι είναι η στάση σωστή και αυτή θα είναι η στάση που θα κρατήσουμε και αύριο το πρωί στην ψηφοφορία. Όταν μιλάμε τώρα για διαδικασίε. έχω την εντύπωση ότι εδώ στο Κοινοβούλιο έχουν γεννηθεί πάρα πολλέ προσδοκίε σε σχέση με αυτό το φάκελο. Είναι σημαντικό φυσικά θέμα, αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν την απόψη τους. Ευτυχώς η στάση της Κομισιόν είναι γνωστή και σαφής. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μας θα ήταν να ξέρουμε και ποια είναι η στάση του Συμβουλίου σε σχέση με το ρόλο του ρυθμιστή. Ξέρω ότι ορισμένοι μας λένε από το Συμβούλιο ότι λένε ότι μπορούμε να συζητήσουμε για τους ρυθμιστές τα επόμενα πέντε χρόνια. Όχι, αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αποτελεσματικές τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ τα κράτη-μέλη προσπαθούν να τροχοπεδίσουν τη διαδικασία αυτή εξυγχρονισμού. Αυτό όμως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μια σαφή έκκληση προς την Προεδρία του Συμβουλίου να προχωρήσει τα πράγματα. Ο κ. Κράμερ αναφέρθηκε και από το κόστος το οποίο δεν καταλογίζεται. Ίσως δεν θυμάται ότι το θέμα των ε, παιδικών σταθμών και των υπηαγωγείων το έχουμε διαγράψει, οπότε δεν είναι πια ένα θέμα. Και επίσης θέλουμε να προσθέσουμε ότι θέλουμε μια σωστή, ένα σωστό διαχωρισμό μεταξύ των ε, υποδομών και της λειτουργικότητας. Αλλά έχουμε πολλές περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, άμα το φέρουμε αυτό σε ακραίο σημείο, όταν γίνεται ένα ατύχημα και δεν μπορεί η εταιρεία που λειτουργεί το, σιδηρόδρομο να έχει επαφή με αυτούς που έχουν τις υποδομές, αυτό δεν είναι θετικό. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το έγγραφο αυτό με πιο πραγματιστικό τρόπο μέχρι να φτάσουμε στην Ολομέλεια. Κύριε Γκρός, μέχρι τις 5 απόψε το βράδυ να ανοιχτεί η προθεσμή για τις προφορικές ε, τροποποίηση της τροπολογίας. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκρός. Πρέπει να αποφύγουμε να καταθέσουμε επιπλέον τροπολογίες. Μέχρι τις 5 έχουμε προθεσμία, αλλά θα μπορούσαμε να καταθέσουμε προφορικές τροπολογίες. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό είναι να ψηφίσουμε, να δούμε πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και να δώσουμε μία σαφή θέση του Κοινοβουλίου. Τώρα σε μια επόμενη φάση μπορούμε να ετοιμάσουμε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και θα αποφασίσουμε τότε για το τι πραγματικά θεωρούμε σημαντικό ενίσχυση του ρόλου του ρυθμιστή, την δημιουργία ενός Ευρωπαίου ρυθμιστή, παρά, τις παραγράφους που αφορούν στην ενίσχυση της διαφάνειας. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να θέσουμε τους διάφορους ε, λειτουργούς ε, του κλάδου σε ισοτιμία. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια διότι άκουσε πάρα πολλές κριτικές στο παρελθόν και σήμερα όλοι την επενούν γιατί κατάφερε να βρει μια συνένεση σε ένα θέμα πάρα πολύ πολύπλοκο. Χρειάστηκε τελικά να συνδυάσει το ασυνδύαστο. Κυρίως όσον αφορά στο θέμα του διαχωρισμού μεταξύ παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης υποδομής. Η Κομισιόν θα πρέπει να το ξανασκεφτεί το θέμα και θα επανέλθουμε όταν θα συζητήσουμε για το θέμα της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και της απελευθέρωσης των εθνικών σιδηροδρομικών φορέων. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να παραμείνει αυτός που παρέχει την υπηρεσία και να συνεχίζεται να χρηματοδοτείται. Πρέπει να παραμείνει το δικαίωμα της απεργίας, οι κοινωνικές πτυχές έχουν συμπεριληφθεί και αυτά ήταν τα στοιχεία που ήταν ενδιαφέροντα για την ομάδα μας. Προσπαθήσω να είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Όλοι ξέρουμε ότι το πρώτο πακέτο για τους ιδεοδρόμους δεν εφαρμόστηκε πλήρως και ξέρουμε ότι ακόμα χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις στα σιδηροδρομικά στην Ευρώπη. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να βρούμε μια σειρά από συμβαστικές λύσεις. Η κυρία Σερακιάν το κατάφερε. Τρίτο σημείο, είπαμε ότι χρειαζόμαστε εθνικούς ρυθμιστές, συμφωνούμε όλοι, αλλά θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε την αποδεσμοποίηση αργότερα Έχουμε ακόμα το 6-4 στο κείμενο και μέχρι τελευταία στιγμή ερχόντουσαν και νέες διατυπώσεις για το άρθρο 6 παράγραφος 4. Αλλά, εν περιπτώσει, θα ψηφίσουμε. Και για τους φιλελευθέρους και για τα θέματα αυτά των παιδικών σταθμών, νομίζω ότι είναι ακόμα μέσα στους υπολογισμούς αυτούς τιμών. Θα πρέπει να σκεφτεί λοιπόν αν από τους παιδικούς σταθμούς και την, νηπιαγωγία εξαρτάται η κερδοφορία και η βιωσιμότητα των υπηρεσιών. Το σκέφτεται αυτό το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Βαντάλε για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν μου φάνηκε να κατάλαβα ότι ο συνάδελφος Δρεμόσα μπορεί να πιστεί με τα πλέον εκτίματα της διαχείρισης της ενωτικής διαχείρισης πέρασαν, έγινε αυτό στη χώρα μου και ήταν πολύ θετικά όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν εμείς να υποστηρίξουμε το διαχωρισμό. Δεύτερο, βλέπετε κύριε Πρόεδρε πόσο ογκώδες ήταν αυτό το πακέτο. Χρειάστηκε να κόψουμε ένα σωρό δέντρα για να καταλήξουμε σε αυτόν τον συμβιβασμό. Ελπίζω στο τέλος της ψηφοφορίας να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Θα είναι σαφείς οι αποφάσεις που λάβαμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν στο τέλος της ψηφοφορίας η συγγήτρια να μας κάνει μία περίληψη των όσων ψηφίσαμε. Και επίσης κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό τον τεράστιο τόμο διότι έχουμε όλο αυτό το χαρτομάνι είναι μια χωριστή λίστα ψηφοφορίας γερμανική. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να ξανακαθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε. Και μετά την ψηφοφορία, θα ήθελα δηλαδή αύριο, να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς κάναμε και να το καταλάβουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μπακ. Νομίζω ότι η νέα διατύπωση αυτού του πακέτου ήταν φυσικά ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και προφανώς θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους άλλους εμπλεκομένους στις διαπραγματεύσεις για τα αποτελέσματα που μπορέσαν να εξασφαλίσουν σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι μπορέσαμε να ξεπεράσουμε πολλά σημεία ασάφεια με αυτέ τι διαπραγματεύσει. Επειδή οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν θίξει τα σημεία που ήθελα και εγώ αναφέρω, θα περιοριστώ σε δύο-τρία μονάχα. Θέλω ιδιαίτερα να υποστηρίξω το γεγονός ότι η κοινωνική διάσταση βρήκε μια θέση σε αυτό το, το φάκελο και δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω γιατί υπάρχουν ορισμένοι μεταξύ μας που θέτουν ένα αμφιβόλο τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για τον ανταγωνισμό επίσης είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρξει μια πραγματική ανεκτή αγορά όταν υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων μεταφορέων και γι' αυτό έχω δυσκολία με την ε, τροπολογία συμβαστική H για την ε, εσωτερικοποίηση των, ε, του κόστους διεθνής, διεθνών μεταφορών. Επίσης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και κάποιο, κάποιος ανεξάρτητος φορέας ο οποίος γιατί δεν μπορούμε με τον τρόπο αυτό να δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να εξασφαλίσουμε την, ε, την ισότητα ανταγωνισμού στο θέμα αυτό. Θα πρέπει με το νομοθετικό αυτό κείμενο να είμαστε ρεαλιστέ. Προφανώ δεν θα επιληθούν όλα τα προβλήματα τα οποία βρισκόνται ενώπιον μα. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πρέπει ακόμα να ρυθμίσουμε στον τομέα των ε, μεταφορών με σιδηρόδρομο. Χρειάζεται νέες, χρειάζονται νέε επενδύσεις στις υποδομές και στα υλικά, μια α, απλοποίηση των κανόνων και επίση, βλέπουμε πολλέ φορέ ότι κλείνουν σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταματούν να λειτουργούν σταθμοί. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε το, την ανάγκη να, ε, να εξυπηρετεί το καταναλωτής και όχι να παίρνουμε αποφάσεις μονάχα ε, ιδεολογικά. Δύο λεπτά κυρία Γιάλα Σέντερ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Σιρακιάνη, όπως επίσης και τους και ε, επίσης, ε, εγώ συμμερίζομαι την άποψη της εισηγήτριας σχετικά με το να κρατήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την χρηματοδότηση των υποδομών ε, και να τους κρατήσουμε χωριστά από τους που παρέχουν την υπηρεσία. Να πω στον κύριο Κράμερ ότι όταν μιλάει για την Ισπανία και θεωρώντας δεδομένο ότι εμείς ε, ξεχωρίσαμε, κάναμε το διαχωρισμό και ότι αυτός ο διαχωρισμός ε, δεν άνοιξε τις μεταφορές. Ε, ξέρετε, εμείς έχουμε τα Πυρηναία, θέλω να ξέρω από πού θα περάσουν αυτά τα τρένα για να μπορέσουν να έχουμε μεγαλύτερη απολευθέρωση ε, της αγοράς στην Ισπανία. για το θέμα της ε, ανοιχτής πρόσβασης ε, στους ε, επιβάτες. Το είπε και το Κοινοβούλιο ότι δεν είναι η ώρα. Ξέρετε από τη χώρα σας ότι ένα holding κάλλιστα μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί όποτε θέλει η χώρα σας έχει την εμπειρία εγώ πιστεύω ότι μπορούμε μέσα από τον ρυθμιστικό οργανισμό να ξεπεράσουμε αυτή την, ε, αυτή τη λογική του holding και όταν θα έχουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να είμαστε εξασφαλισμένοι. Θέλω να έχουμε ισχυρούς εθνικούς ρυθμιστές και ελπίζω να μπορέσουν να καταφέρουν να προχωρήσουν όλες ε, τις συστάσεις που θα τους δώσουμε για να, προχωράσουμε, να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή σιδηροδρομική ολοκλήρωση όπου δεν θα έχουμε holdings ευνοούμενα έναντι άλλων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα. Διαπιστώνω πόσο ήταν πολύ σημαντική αυτή η αναβολή. Ε, πρόκειται εδώ για μια φιλική αναθεώρηση των ρυθμίσεων. Θεωρώ όμως ότι είναι ανεπαρκές. Το τρίτο σημειώνουμε τις επιθυμίες που εκφράζει η Κομισιόν του χρόνου να μας δώσει μία βάση εργασίας για τον διαχωρισμό και το άνοιγμα των αγορών. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το ένα χωρίς το άλλο. Δύο παρατηρήσεις. Εγώ περιμένω να δούμε τι θα μας πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Βέβαια δεν, θέλω να είναι ο δικαστής να είναι ή ε, ο νομοθέτης να είναι αυτός που ακούει τι του λέει ο δικαστής. Ε, θέλω ο δικαστής να ακούσει τι θα του πει ο νομοθέτης. Πάντως εμείς εδώ είμαστε πραγματικά ο τελευταίος χώρος που έχει απομείνει που συζητάμε τον διαχωρισμό μεταξύ της διαχείρισης της υποδομής και της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς. Διότι παντού έχει λυθεί. Η κατσίκα του κύριου Σεγγέν, ένα διήγημα, γράφτηκε τον 19ο αιώνα, είναι πάρα πολύ γνωστό και η κατσίκα του κυρίου Σεγγέν έφυγε στο βουνό για να ε, γευτεί την ελευθερία της και έπεσε πάνω στο λύκο το βράδυ ε, και ε, το, βράδυ έφτασε ο λύκος, πολέμησε με το λύκο όλη τη νύχτα για να επιζήσει, αλλά το πρωί ο λύκος την έφαγε. Ποιο είναι ο λύκο τώρα στου σιδηροδρόμου, θα ήθελα πολύ να ξέρω. Κύριε Τικάου, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία Σερακιανή, η οποία εργάστηκε πάρα πολύ και αξίζει όλες τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι η ανάπτυξη των υποδομών στο σιδηροδρομικό τομέα θα πρέπει να προχωρήσει και αφού έχω μιλήσει με όλους τους εμπλεκομένους, με τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους των ε, χρηστών, βλέπω ότι αυτή η στρατηγική είναι πολύ θετική. Είχαμε πολλές συζητήσεις αλλά δεν έχουμε αναφερθεί πάρα πολύ ούτε στους ε, καταναλωτές ούτε στα συνδικάτα. Κατέθεσα την τροπολογία 357 στο σημείο στην παράγραφο 9 και ζήτησα να διαγραφεί η τροπολογία αυτή που έχει να κάνει με το χρέος των θηγατρικών εταιριών. Οι θηγατρικές πολλές φορές όμως έχουν χρέη προς τις τοπικές αρχές. Είναι χρέη τα οποία έχουν προξενηθεί από κοινωνικέ υποχρεώσει. Θα ήταν κατά την άποψή μου σφάλμα να μην λάβουμε υπόψη αυτή την πτυχή και επομένω να διαγράψουμε το χρέο των θεατικών αυτών επιχειρήσεων. <clears throat> Επίση σημαντικό είναι να αποδεχθούμε το γεγονός ότι όταν μιλάμε για την πρόσβαση στις υποδομές σιδηροδρομικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να είναι αδύνατο οι επιβάτες να παίρνουν πληροφορίες για τα θέματα αυτά. Και να είναι πολύ δύσκολο να αγοράσουν ένα εισιτήριο για να πάνε από το α στο β. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν να αξιολογήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εργατικό δυναμικό και οι κοινωνικές ε, συνθήκες και πώς προχωράει η εξέλιξη των συνδρομικών συγκοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει επίσης και μια τροπολογία R, λατινικό, που αφορά το σημείο 8. Δεν πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να επιδοτούμε τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περάσει στο σύστημα RTS, δηλαδή για την αυτόματη, για την αυτόματη σηματοδότηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε τις πιο μεγάλες εταιρείες και όχι αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ε, επενδύσει σε αυτά τα συστήματα. Όχι, όμως πρέπει και οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να έχουν το χρόνο να προχωρήσουν προς ένα εξυγχρονισμό των συστημάτων τους. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε για μια μείωση για αυτούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε τέτοιες επενδύσεις. κ. Πάκερ για την Κομισιόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ την εισηγητρία για την εξαιρετική εργασία της. Υπάρχει μια βάση για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Η Κομισιόν είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη, συναφώς. Πρόεδρε, να σχολιάσω κάποιες από τις τροπολογίες, όχι όλες, για να σας πω πώς τις βλέπουμε. Πολλές από τις τροπολογίε συνάδουν με την σχέση με την θέση της Κομισιόν. Κάπου αλλού έχουμε αιτήσει για διευκρινήσεις, θα σας τις δώσουμε. Στις συμβαστικές τροπολογίες ουσιαστικά ενισχύεται η θέση της Κομισιόν. Γενικά είμαστε υπέρ αυτών των τροπολογιών, με τις οποίες εν γέννη παρατείνεται η ισχύ των εθνικών διατάξεων μειώνονται οι προθεσμίες για να κλείσουν οι συλλογισμοί των εταιριών λειτουργίας, τροποποιούνται τα χρέη, τα τέλη χρήσης δικτύου σε αρτήση του προκαλμένου θορύβου, τροποποιούνται ορισμένες, τρο... ορισμένες προθεσμίες και το μόνο που ήθελα να σημειώσω εδώ είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την ιδιαίτερη διατύπωση αυτών των τροπολογιών, ώστε να μην προκληθεί επιπλέον περιττή γραφειοκρατία τόσο για τι εταιρείε όσο και για του δημόσιου τομεί και για την Κομισιόν και για να αποφύγουμε τι αρνητικέ επιπτώσει στην αγορά. Κατά άλλα, θα βελτιώσουμε το κείμενο όσο μπορούμε. Κάποιε τροπολογίε, όπω είπα, συνάδουν με τη θέση των ε, νομικών είναι το άρθρο 13, μια βασική ρήτρα, μια βασική διάταξη όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο. Η πρόταση αυτή είναι κάτω από την αρχική πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά την υποχρέωση αποδέσμευσης. Εκφράζω πίστη την ικανοποίησή μου για την πρόθεση του εισηγητή να ευνοήσει τη δεύτερη ανάγνωση. Πρόεδρε, υπάρχουν λίγες τροπολογίες οι οποίες είναι κάτι από αυτό το οποίο θα ήθελε να πετύχει η νομική υπηρεσία που δημιουργούν παραθυράκια. Υπάρχουν δηλαδή τροπολογίες οι οποίες μας γεννούν ανησυχίες και τροπολογίες που δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε. Η πιο σημαντική, να την αναφέρω, είναι αυτή η οποία αναφέρεται στον υπολογισμό των αμέσων στοιχείων του κόστους. Παράδειγμα 8, στοιχείο 1. Υποχρέωση των διαχειριστών υποδομή όταν αξιολογούν τη δυνατότητα χρέωσης περιθωρίου κέρδου. Οι ρυθμιστικέ αρχές οι οποίες ε, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην περίπτωση ανεπιθυμητών εξελίξεων στο 56 και το θέμα του αντικειμένου των εκχωρημένων αρμοδιοτήτων. Όλα αυτά, αν θέλετε, τα βλέπει η Κομισιόν πιο απειρητικά και πιο φιλόδοξα. Υπήρχαν και ερωτήσει, ε, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά συγκεκριμένε τροπολογίε. Αν θέλετε, μπορώ να αναφερθώ και σε αυτέ. Να ξεκινήσω από την 357, κύριο Κάου, όσον αφορά τα χρέη, τα προηγούμενα χρέη. Έχουμε ξεχωρίσει, έχουμε αποκλείσει, έχουμε εξαιρέσει τις θεατρικές, γιατί είτε είναι συνδυασμικές επιχειρήσεις, που είναι θεατρικέ των μεγάλων εθνικών οργανισμών σιδηροδρόμων ε, είτε δεν υπάρχει λόγος από την άλλη μεριά να τους δώσουμε ειδική ενίσχυση βάσει των κανονών περιθνικών ενισχύσεων. Άρα και αυτή η διάταξη παραμένει. Τώρα, όσον αφορά την προφορική τροπολογία 2, άρθρο 2, κ. Μαρινέσκου, την οποία υποστηρίζουν και άλλοι, αν δεν κάνω λάθος, επέκταση της ε, εξαίρεση του γύρω τάνελ όσον αφορά τους κανόνες χρέωσης. Είναι αρκετά πολύπλοκο το ζήτημα και ανησυχεί και την Κομισιόν. Σήμερα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί μπορεί να εξαιρεθεί από τους κανόνες, αλλά υπάρχουν ελάχιστε απαιτήσει που πρέπει να διατηρηθούν. Οι διαχειριστέ υποδομών δηλαδή πρέπει να χρεώνουν βάση του μακροπρόθεσμου κόστους. Σας ενημερώνω επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε διαδικασία επί παραβάση κατά της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ακριβώς σε σχέση με τον κύριο Τάνελ επειδή δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ της υποδομής και των χρεώσεων. Είναι κομμάτι του σιδηροδρομικού και εκτιμένου αν θέλετε. Και λίγα λόγια για την τροπολογία το ε, στο 26, αρχικός προφορική τροπολογία, τώρα περιλαμβάνεται στην τροπολογία συμβαστική A, σχετικά με τη μεταφορά πόρων από το διαχειριστή της υποδομής προς το holding. Πρέπει το κεφάλαιο αυτό να ε, αποπληρώνεται με κάποιο τρόπο. Μπορεί να φαίνεται απλό και λογικό, αλλά είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, η ρυθμιστική αρχή να επιβάλλει αυτόν τον κανόνα εάν δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία. Εδώ με την προσοχή της Επιτροπής σας όσον αφορά αυτή την συμβαστική τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία 4 στο άρθρο 10 του κ. Τρεμόζα. Είναι πολύ απλή. Εσείς λέτε να διαγράψουμε τη λέξη διεθνής, international. Και έτσι να ανοίξουμε πιο γρήγορα τα σύνορα στι εσωτερικέ μεταφορέ επιβατών. Δεν ήταν αυτό ο στόχο, αλλά ακόμη και το άρθρο αυτό δεν θα αρκούσε για να γίνει αυτό στην πράξη. Άλλωστε, θα συμφωνήσετε, χρειάζεται προετοιμασία ε, στο δεύτερο εξάμεινο του 12 για να μπορέσουν τέτοιε προτάσει να υποβληθούν και να μελετηθούν. Για να ανοίξει δηλαδή και η εσωτερική κυκλοφορία ε, μεταφορά μάλλον επιβατών. 7 στο άρθρο 31 διαφοροποιούμενα τέλη χρήση υποδομών με δημόσια χρηματοδότηση. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω ε, αν ε, η αναδιατύπωση αυτή είναι κατάλληλη ευκαιρία να περάσουμε αυτή την ιδέα, αλλά το ότι μπορούν να διαφοροποιούνται, να διαφοροποιούνται οι χρεώσει βάσει τη χρηματοδότηση και τη συναρτήσει του προκαλουμένου θορύβου είναι μια ιδέα που βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μάλιστα, θέλει ότι με τον χρηματοδοτικό μηχανισμό Connecting Europe που θα δρομολογηθεί σε λίγε μέρε, έχουμε έναν εξαιρετικό τρόπο να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα μείωση του θορύβου στα κράτη-μέλη. Ίσως εκεί θα ήταν καλύτερο να δούμε το θέμα. Και να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με μια τελευταία παρατήρηση. Είναι παλιά πρόταση της Κομισιόν. Υπάρχουν τροπολογίες στο άρθρο 4 και στο 19, στο 21, 27, 52 και 57. Και 54, με συγχωρείτε. η πρόταση αναδιατύπωση δεν τροποποιεί αυτέ τι διατάξει. Οπότε, θεωρώ, κατά τη δική μα ερμηνεία, σύμφωνα δηλαδή με του κανόνε τη αναδιατύπωση, ότι εν γέννη αυτές οι διατάξει δεν πρέπει να τροποποιηθούν ουσιοδό. Εκτό αν πρόκειται για λόγου αυτοσυνέπειε του κειμένου. Αλλά δεν μπορούν να τροποποιηθούν, επαναλαμβάνω, επί τη ουσία. Αυτό το γνωρίζετε, κύριε ε, Πρόεδρε, θα σα το επιβεβαιώσω και γραπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σε σχέση με την τελευταία σας παρατήρηση, το καταγράφουμε αυτό το οποίο λέτε. Φυσικά είναι κυρία το Κοινοβούλιο για να αποφασίσει. Κυρία Σερακιάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά σύντομα. Διότι μερικά τα ξεκαθάρισε η Κομισιόν και άλλα τα ξεκαθάρισαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας διασφαλίσω ότι η εργασία μας ήταν ιδιαίτερα συνεργατική. Ευχαριστώ τους και όδης εισηγητές και φυσικά δεν είχε πρόθεση αυτή η συνεργασία να χειροτερεύσει το κείμενο του πρώτου συνδυνοδρομικού πακέτου διότι δύσκολο εξάλλου θα ήταν να κάνουμε χειρότερα από ό,τι είχε γίνει μέχρι τώρα διότι το πρώτο τμήμα δεν είχε εφαρμοστεί και για το υπόλοιπο είχαμε 17 διαδικασίες παραβίασης, 4 λιμένες και 13 εκκρεμούσες. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα τέλειο κείμενο, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει και ένα τέλειο κείμενο. Σίγουρα θα χρειαζόταν μεγαλύτερη φιλοδοξία εκ μέρους της Κομισιόν που είχε αλλάξει και θέση κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Τώρα όμως μεσολαβεί η πιο δεσμευτική φάση των εργασιών μας να κρατήσουμε και ορισμένα σημεία του κειμένου στα οποία ε, το Κοινοβούλιο πραγματικά μετράει τον ε, ρυθμιστή, το θέμα της χρηματοδότησης των υποδομών, το κόστος ε, και όσα γράφονται ως δεσμεύσεις στα άρθρα 6 και 7 και τα οποία ζητάμε από την Κομισιόν. Αυτή θα είναι η πιο σκληρή δουλειά. Αύριο είναι πολύ πλοκή η ψηφοφορία. Θα έχουμε και το απόγευμα μια νέα voting list, διότι ελέγχοντας είδαμε ότι είχαμε δύο-τρία λάθη. Θα ξανασταλεί η voting list, παρακαλώ να την ξαναελέγξετε, διότι ο μέγας αριθμός τόσο τροπολογιών και συμβιβασμών σίγουρα κάποιο λάθος μπορεί να μας ξέφυγε ο κατάλογος ψηφοφορίας έχει γίνει και αν περάσουν φυσικά οι συμβιβασμοί το κείμενο είναι συμβατό. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί φυσικά θα αλλάξει και το κείμενο και τότε θα το συζητήσουμε στο τέλος της ψηφοφορίας. Τώρα σχετικά για την απεργία. Ξαναλέω ότι το αφήσαμε απ' έξω και λάβαμε υπόψη μας ότι σαφώς τα κράτη-μέλη ε, και αλλού λιγότερο σαφώς έχουν την αρμοδιότητα. Τώρα για το ποιος είναι ο λύκος ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είναι, μπορώ να σας το πω. Αλλά όχι εδώ, αλλού να σας το πω. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό κύριε Σερακιάνη. Επειδή είπατε για την ψηφορία είναι αύριο. Έχουμε ένα κατάλογο ψηφορία, τρένο ολόκληρο που με κόπο φτιάξαμε αυτήν την εβδομάδα Ενώψη ώψη τη επόμενη συνόδου τον Νοέμβριο. Αύριο λοιπόν είναι 6.40, μην ξεχάσετε τι κάρτε σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σερακιάν. Το επόμενο σημείο είναι η τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα. Λάβετε θέσεις. Εισηγητής, κύριος Φλέκενστάιν. Όσοι να φύγουν παρακαλώ ήσυχα και αν έχετε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 Τι ωραία που όταν συζητούμε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα όλοι εγκαταλείπουν το πλοίο. As ever, the Commission is noisiest section at the moment. Can you? Λίγη ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά. Χρειάζομαι ησυχία, διότι πριν ακούσουμε τον κύριο Φλέκενστάιν, πρέπει να καλωσορίσω για τελευταία φορά τον κύριο Βιμτερόιτε, ο οποίος είναι ο προχώμενος πρόεδρος της ΕΜΣΑ, ο οποίος σε λίγο δεν θα είναι εκεί πλέον. Διορίστηκε το 2003 στην θέση αυτή. Τον γνωρίζουμε, βεβαίω και προηγουμένω ήδη εργαζόταν στην Κομισιόν πριν την ΕΜΣΑ. Ήθελα πάντω να πω ότι διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη δημιουργία στην οικοδόμηση τη ΕΜΣΑ. Θα ήθελα και προσωπικώ να τον ευχαριστήσω για τα όσα έκανε. Αλλά είμαι βέβαιο ότι απηχώ τι ευχέ όλων σα για την καλή συνταξιοδότηση και τα όλα όσα έχει να κάνει από εδώ και πέρα. Κύριε Βεντερόη, ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σα κάνουμε τη ζωή δύσκολη τελευταία φορά που έρχεστε εδώ. Ο κύριο Φλέκενστάιν έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τους και όλους και δεν το λέω μόνο από ρητορία ή συνήθεια, απλώς είμαι πεπισμένος ότι καταφέραμε να συνεργαστούμε μια χαρά. Εμείς εξεργαστήκαμε συμβιβασμούς φυσικά όταν έχουμε συμβιβασμούς δεν μπορεί να πετύχει ο καθένας να έχει όλα όσα θέλει για μένα υπάρχουν σημεία που σίγουρα θα ήθελα να έχουμε περισσότερα ε, αλλά αυτά που πετύχαμε μας όφελ, μας βοηθούν να έχουμε μία επαρκή πλειοψηφία για να πάμε να συζητήσουμε έγκυρα με το Συμβούλιο. Και αύριο θα ζητήσω την εντολή σας ε, για να μου πείτε εάν μπορώ να διαπραγματευτώ ή όχι. Εγώ έψαξα να δω κατά πόσο εδώ επέφταμε σε αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ ή επρόκειτο για κάτι το καινούριο για να μην υπάρχει επικάλυψη με, τους, με, τις, δραστηριότητες της ΕΜΣΑ για να μπορέσουμε να έχουμε πάντοτε προστιθέμενη αξία σε όλες αυτές τις πράξεις και να έχουμε και τη σωστή ισορροπία μεταξύ κόστους ωφέλειας. Κάποιες παρατηρησούλες ακόμα. Έχουμε ήδη ασχοληθεί στο θέμα αυτό των υπερακτίων δραστηριοτήτων σε σχέση με την ασφάλεια στη θάλασσα. Έχουμε πάντα τις ε, αιτήσει των κρατών μελών και της Κομισιόν, ε, μάλλον τη συνεισφορά των κρατών μελών και της Κομισιόν που ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Ένας ενιαίος θαλάσσιος χώρος χωρίς σύνορα είναι μια άποψη, όπου, είναι μια αντιμετώπιση όπου η ΕΜΣΑ ή η ΕΟΑΘ θα μπορούσε σίγουρα να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εδραίωση αυτού του ενιαίου χώρου. Ξέρουμε ότι τα θέματα τα θαλάσσια είναι πολύ σημαντικά και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ο ΕΟΑΘ, ΕΜΣΑ, στο βαθμό που σε σημαντικούς τομείς όπως είναι η κατάρτιση των ναυτικών ε, δεν μπορούν βέβαια να αναλυφθούν από αυτόν τον οργανισμό, δεν μπορεί να γίνει εκπαιδευτής ναυτικών η ΕΜΣΑ, αλλά βάσει της παγκόσμιας ε, εμπειρία μας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μεταλαμπάδευση βελτίστων εμπειριών και σε διεθνείς επαφές και μπορεί να γίνει αυτό με πιο πρόσφορο τρόπο μέσα στα πλαίσια ενός δικτύου της ΕΜΣΑ και με άλλους ε, οργανισμούς. Το θέμα της πειρατείας επίσης είναι κάτι το οποίο από, στο οποίο από μόνη της η δράση μας ήταν εύγλωτη. Υπάρχουν τρία θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μένα και τα οποία δεν καλύπτονται στις συμβιβαστικές θέσεις. Έχουμε συζητήσει καταρχήν για τα μέτρα διάσωσης, για το αν θα πρέπει να περιληφθούν στις αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ ή όχι. Κατά τη δική μου άποψη, τα σωστικά μέσα και οι σωστικές δραστηριότητες βρίσκονται ήδη και σήμερα μέσα στις αρμοδιότητές της και όταν μιλάμε με την, με την ε, νέα αντιμετώπιση της διάσωσης, δηλαδή στην ανοιχτή θάλασσα, στην, ε, με χρήση ελικοπτέρων και άλλων ε, εξοπλισμών. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό, αλλά τουλάχιστον η τωρινή αρμοδιότητα που έχει σε παράκτια διάσωση θα πρέπει να παραμείνει. Ένα τρίτο θέμα είναι η συζήτηση του κατά πόσο θα είναι οι εθνικές ή <clears throat> περιφερειακές αρχές οι οποίες συνεργάζονται με την ΕΜΣΑ και η δική μας άποψη ήταν στις συμβαστικές τροπολογίες ότι πρέπει να είναι εθνικές αρχές, γιατί οι περισσότερες αρχές είναι εθνικές, αλλά όταν υπάρχουν ήδη κατανεμημένες αρμοδιότητες σε περιφερειακό επίπεδο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουν αυτές την αρμοδιότητά τους. Και ένα τελευταίο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι η πολιτική φύλου. Στο Κοινοβούλιο έχουμε καταλήξει σε ένα σαφές ψήφισμα στη θέση που δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω, αλλά πρέπει και για την ΕΜΣΑ και για άλλους φορείς να είμαστε σαφείς ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και ότι έχουν την ευθύνη της ε, εφαρμογής τους και στην πράξη. Συνολικά όμως νομίζω ότι η συνεργασία μας είναι το απάβγασμα μιας γενικής εντύπωσης ότι λειτουργεί πολύ καλά η ΕΜΣΑ. Και θέλω να ευχαριστήσω την, ε, την, ε, τους εκπροσώπους της ΕΜΣΑ για τη συνεργασία τους και για ε, τη βοήθεια που μας έχουν δώσει στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και τον εισηγητή. Πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Φλέκενσταν, η διάθεσή σας για συνεργασία κτλ. Και εμείς ήδη θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή η έκθεσή σας. Το κείμενο της Κομισιόν βέβαια ήταν φιλόδοξο, δεν πρόκειται εγώ να το επικρίνω. Μέχρι τη στιγμή Μέχρι τώρα η ΕΜΣΑ ήταν ένα υποδειγμα, ένας υποδειγματικός φορέας ο οποίος έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντερόιτερ γιατί μέχρι τώρα ήταν πραγματικά υποδειγματική η εργασία του. Τώρα, το θέμα είναι το θέμα των ε, αρμοδιοτήτων, το θέμα του οργανογράμματος της ε, ΕΜΣΑ, η συνεργασία με γειτονικές χώρες και η αντιμετώπιση των πλατφορμών εξόριξης πετρελαίου στην ανοιχτή θάλασσα για να αντιμετωπιστούν τα θέματα ρήπανση. Μετά από το ατύχημα του κόλπου του Μεξικού είναι φανερό ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερε αρμοδιότητε στα θέματα αντιμετώπιση τη ρήπανση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε στον εισηγητή όλοι μαζί μια εντολή που θα εξασφαλίσει την συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Το έγγραφο του εισηγητή είναι εξισορροπημένο, δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ΕΜΣΑ αλλά εγώ θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες δικές μας που θα τις παρουσιάσω τηλεγραφικά. Στο ΕΛΚ για τις αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ υπάρχει συνένεση ότι πρέπει να αντιμετωπίζει η ΕΜΣΑ τα θέματα της ασφάλειας στη θάλασσα. Και έχουμε διατυπώσει και μια τροπολογία συμβαστική, την τροπολογία 2 εισηγητής, με την οποία συμφωνούμε. Και άλλες πολιτικές ομάδες συμμετέχουν σε αυτή την συμβαστική λύση. Δεύτερον, εγώ υποστηρίζω την, ε, το συνδυασμό της ΕΜΣΑ με άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και την μεταλαμπάθευση βελτίστων πρακτικών. Οι υπηρεσίε ακτοφυλακής, το τρίτο θέμα. Εμεί θέλουμε να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών που ελέγχουν τις παράκτιες περιοχές. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και είμαστε κατά της τροπολογίας συμβασμού 4 σε σχέση με τον πολλαπλασιασμό των ε, κέντρων εκπαίδευση που θα μπορούσε να είναι κάτι το περιττό. <coughs> Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προωθήσουμε το ναυτικό επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό υποστηρίζουμε την προφορική τροπολογία Α και τη συμβασική τροπολογία 3. Επίσης, υποστηρίζουμε να υπάρξει, όπως ζητούν οι τροπολογίες 98 και 99, να υπάρξει βοήθεια από την ε, ΕΜΣΑ, τα κράτη-μέλη και τι περιφερειακές αρχέ για τη σύλληψη σκαφών που προσπαθούν να διαφύγουν τη δίωξη. Υποστηρίζουμε λοιπόν όλε τι συμβαστικέ τροπολογίε εκτό από τι θέσει και τέλο για την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Μου φαίνεται πολύ καλή συμβαστική λύση 6, η οποία περιλαμβάνει μια σύσταση στον τομέα αυτό. Θεωρούμε όμω ότι τώρα επιβάλλουμε μια υποχρέωση. <coughs> Όπω ζητείται από την προφορική ερώτηση ε, τροπολογία Δέλτα, αυτό είναι υπερβολικό. Είναι άλλο μια σύσταση και άλλο μια υποχρέωση για την ε, ισότητα των φύλων σε επίπεδο. Επίσης το ΕΛΚ έθεσε τις τροπολογίες 90 βλάστο κερκές και την 98 Κανθεάν 172 του κ. Κουμουτσάκου. Όλες αυτές τις τροπολογίες υποστηρίζουμε και ελπίζουμε ότι θα ευδοκιμήσουμε. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συναδέλφους που με άφησαν να μιλήσω εξ ονοματός τους μετά από μια αγαστή συνένεση και με άφησαν να εκπροσωπήσω τη θέση του ΕΛ προς τους συναδέλφους. Για τις τροπολογίες του, του, της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Περιβάλλοντος υποστηρίζω τις συμβαστικές θέσεις του εισηγητή και ελπίζω ότι αύριο θα είναι θετική όπως το απαιτεί και το έργο του εισηγητή και των άλλων μελών της Επιτροπής. Thank you very much. Now, Mrs. Bilbao for the... Ευχαριστώ κύριε για τους Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω προφανώς ευχαριστώντας τον εισηγητή, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία. Ένα πάρα πολύ εμπεριστατωμένο έργο. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία ελέγχθηκαν ήδη από τους προλαλήσαντες. Θέλω να τονίσω ότι συμφωνούμε, όπως είπαμε και προηγούμενα, με όλες τις συμβαστικές τροπολογίες εκτός από την υπαριθμόν 6 που αφορά στη συμμετοχή ανθρώπων και γυναικών. Ακούσαμε μόλις τον κύριο Ντεπασκουάλ που λέει ότι και το ΕΛΚ είναι εναντίον αυτής της τροπολογίας. Η συμβαστική τροπολογία εδώ αφαιρεί την ε, ανάγκη να υπάρξει υποχρέωση ισότητος φύλων την φέρνει μοναχα στι αιτιολογικέ σκέψει. Επομένω, αυτό δεν φέρνει κάποια υποχρέωση. Και εξάλλου αυτό δεν είναι κάποιο καπρίτσιο τη ομάδα μα. Εμεί αναφερθήκαμε σε αυτέ τι τροπολογίε, γιατί ήδη τον Ιούλιο το Κοινοβουλίο μα ενέκρινε ένα ψήφισμα <clears throat> όπου υπήρχε υποχρέωση στις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν μια ισότητα ανδρών και γυναικών, μια ισορροπία τουλάχιστον στα διοικητικά του συμβούλια. Δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και το να φέρουμε αυτό το θέμα μονάχα στην αιτιολογική σκέψη, αυτό θα μείωνε την ε, έμφαση για την εξισορρόψη αυτή. Οι άλλες συμβαστικές τροπολογίες πάντως δεν μας δημιουργούν πρόβλημα. Κατά δεύτερο λόγο και μετά από αυτά που είπε και ο ίδιος ο εισηγητής, υπάρχουν τρεις τροπολογίες όπου εμείς θα ζητήσουμε να συμπεριληφθεί κάποια προφορική τροποποίηση 103-61 και η αιτιολογική σκέψη 8, γιατί γίνεται απλώς μια αναφορά της, στην ανασυμπίληση των δεδομένων για τα προσόντα, μια αναφορά στις συνεργίες και όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Εμείς είχαμε τονίσει σε πολλές συνεδριάσεις στο παρελθόν ότι υπάρχουν πολλές φορές και περιφερειακές αρχές οι οποίες έχουν αρμοδιότητες και πρέπει να αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο και προτιμούσαμε να λέγεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή θα μπορούσε να αφήσει κανείς ανοιχτό το θέμα λέγοντας οι αρμόδιες αρχές. Θα διατηρήσουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία γιατί δεν είναι ούτε πολιτικό θέμα ούτε θέμα μονάχα προτίμησης. Είναι ένα θέμα πραγματικών αρμοδιοτήτων και καλύτερης οργάνωσης. Τρίτον, να σας πω ότι θα προτείνουμε μία προφορική τροποποίηση για την τροπολογία 115 για να ενσωματωθεί ένα, μια φράση που αναφέρεται στην ε, έρευνα ώστε να συμπεριληφθεί και η έρευνα για την εξόρυξη σε πλατφόρμες φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Τέλος, για να κλείσω, μπορούμε να ήμασταν θα μπορούσαμε να, είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η συμφωνία η οποία επετεύχθη είναι στα όρια του εφικτού και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αρμόδιοι για πιο φιλόδοξοι για τις αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ για να αποφύγουμε ότι όπως το παρελθόν ανδρώνεται η ΕΜΣΑ μέσα από μια σειρά αποκρίσεις. Χαιρόμαστε που δεν έχει αντιμετωπιστεί το, που έχει αντιμετωπιστεί το θέμα των πλατφορμών για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, για τη δημιουργία του θαλάσσιου χώρου χωρίς σύνορα, για τα θέματα κατάρτισης των ναυτικών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν γίνει δεκτά, γιατί οι περισσότερες ομάδες δεν συμφώνησαν με την ιδέα μιας ευρωπαϊκής σχολής για την εκπαίδευση των ναυτικών, κάτι το οποίο θα είναι προφανώς μια ένα μεγαλύτερο κύρος και ακτινοβολία στο έργο των ναυτικών Επίσης για το θέμα της ε, πειρατείας, νομίζω ότι όλα αυτά ήταν ικανοποιητικά. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία επετέθησαν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ρόιτερ για το έργο του και νομίζω ότι του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ευτυχία στις νέες αρμοδιότητες που θα αναλάβει και ελπίζουμε ότι σε κάποια μετροδική ευκαιρία θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Γιατί τέτοιου είδου θέματα <clears throat> νομίζω ότι είναι θετικά για όλους να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πιο ευρωπαϊκού χαρακτήρα εγχειρήματα όπως αυτό της ΕΜΣ. Ευχαριστώ. Ισία. E e Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισήγητη για την εξαιρετική συνεργασία. Εμείς από την αρχή βλέπαμε κάπως επικριτικά το κείμενο. Ως προς το πώς βλέπουμε την ΕΜΣΑ. Δηλαδή δεν βλέπω να διευρύνουμε έτσι τις αρμοδιότητες ε, της ΕΜΣΑ στον έλεγχο των παρακτήριων περιοχών Αυτό που κάνουν σήμερα τα κράτη-μέλη εμάς μας αρκεί και με το παραπάνω. Είμαστε πιο κοντά λοιπόν με την πρόταση της Κομισιόν. Από την άλλη μεριά υπάρχουν προτάσει εξαιρετικά απαιτητικέ και φιλόδοξες. Δηλαδή δεν βλέπω γιατί εμπλέκουμε την κοινωτική διάσταση σε ορισμένα θέματα να δεν το κάνουμε με άλλα. Υπάρχει επίση ε, μια συμβαστική τροπολογία με την οποία συμφωνούμε όσον αφορά την ε, εμπλοκή της ΕΜΣΑ στην εκπαίδευση ναυτιλωμένων. Τώρα όσον αφορά τη διεύρυνση όμως των αρμοδιορίτων της ΕΜΣΑ, εκεί δεν θα μας βρείτε υποστηρικτές σας. Κύριε Τερότερ, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό. Είμαι βέβαιος ότι σας περιμένουν ευχάριστα χρόνια. Σας εύχομαι υγεία για το μέλλον. Στέλιο για τους πράσινους. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και να ευχαριστώ στον κύριο Φλέκενστάιν για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ σκιωδών με τόση αποτελεσματικότητα. Χαίρομαι που συμπεριλαμβάνονται πλέον οι εξέδρες ε, γεωτρήσεων. Κάτι το οποίο συνάδει με τις ανησυχίες που έχουμε για το περιβάλλον. Επιπλέον, χαίρομαι για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, οργανισμών, με εφαρμογή συγκεκριμένα έργα. Αυτό είναι καλό, διότι αποφεύγονται οι επικαλύψεις. Από την αρχή ήταν ένα από τα πράγματα που με ανησυχούσαν. Ήθελα να ενσωματωθεί δηλαδή αυτή η πρόβλεψη στην δουλειά μας. Θα υποβάλουμε προφορική τροπολογία επί της συμβαστικής τροπολογίας 1. Πρόκειται για θέμα που συζητήσαμε στους σκιώδες όσον αφορά τον ρόλο της ΕΜΣΑ στην παροχή υπηρεσιών διάσωσης, ε, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκη. Είναι μια μικρή προφορική τροπολογία, η την οποία ζητώ την υποστήριξή σα. Ε, προστίθεται δηλαδή η λέξη rescue, ε, διάσωση, στο, στη λέξη assistance, βοήθεια. Ξέρω ότι δεν είναι παντά εύκολα τα πράγματα για τους πρασίνους, αλλά στο πνεύμα της συνεργασίας θα Ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας για αυτήν την μικρή προφορική τοπολογία. Κύριε Μάισνερ. Sorry, μια στιγμή. Κύριο Κόλιτσεκ πρώτα, αν δεν σας πειράζει. Συγγνώμη κύριε Κόλιτσεκ, δεν σας είδα εκεί στη γωνιά. Ήσασταν πολύ αριστερά εκεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Κόλτσεκ. Είμαι μικρός όμως, είμαι πίσω, είμαι αριστερά, όλα αυτά. Αντίθετα τώρα από τους συναδέλφους μου, εγώ δεν έχω μια ιδιαίτερη εμπειρία σε σχέση με τη θάλασσα. Κάνω λίγο κανό, αλλά δεν έχω τόσο στενή σχέση με τη, θάλασσα. Για τις ε, υπεράκτιες εγκαταστάσεις, εξορίξεως κτλ. Εδώ τίθεται ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα <clears throat> και η ΕΜΣΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει καλύτερα ορισμένες πτυχές που είχαμε αναφέρει όταν μιλούσαμε για το κείμενο και το θέμα που είχε να κάνει με τα θαλάσσια ατυχήματα. Υπάρχουν εκεί κοινά στοιχεία, θα πρέπει να μπορέσουμε να, καταλήξουμε σε μια παρόμοια προσέγγιση. Επίσης για την ε, κατάρτιση και την πιστοποίηση των ναυτικών, ακόμα και η τσεχική δημοκρατία που όπως ξέρετε δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, έχει μια σχολή για, το επάγγελμα. Και υπάρχει μια επιτροπή 17 επιτροπών σε, στη χώρα μας και η Επιτροπή του Ρήνου παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαιδευτικών, αμοιβαίας αναγνώριση πιστοποιητικών. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθούν νέες δομές. Υπάρχουν ήδη δομές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα ήθελα του τουλεχθέντο να υποστηρίξω όλε αυτέ τις προσπάθειε οι οποίε έχουν σαν στόχο να πετύχουμε καλύτερο συντονισμό και η ΕΜΣΑ μαζί με την Κομισιόν θα μπορούσαν να συνεργαστούν πιο στενά με την Επιτροπή του Ρήνου η οποία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αμοιβαία αναγνώριση προσόντων. Ευχαριστώ τώρα κύριε Μάσινα. Σας ευχαριστώ. Λίγα σημεία μοναχά χρειάζεται να θίξω γιατί τα περισσότερα τα έχουν πει οι συνάδελφοι και είναι σωστά. Κύριε Πασχουάλ, η, και η ολοκληρωμένη πολιτική της θάλασσας, η έκθεσή μας ανάφερε το θέμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, αλλά δεν το πετύχαμε. Θέλουμε λοιπόν να ε, τονίσουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο ακόμα και αν δεν συμφωνεί η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Για το ναυτικό επάγγελμα ξέρουμε ότι είναι τομέα ανάπτυξης στο ναυτικό επάγγελμα και για τους άνδρες αλλά και για τις γυναίκες και πάρα πολύ ενδιαφέρονται για αυτό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε και περισσότερες σχολές στον τομέα αυτό, όπω είπε και η κυρία Μπιλμπάου. Η εκπαίδευση αυτή λοιπόν για τους άνδρες και τις γυναίκες θα πρέπει να έχει ένα ισότιμο χαρακτήρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι, οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να έχουν διαφορετικές ε, αντιμετωπίσεις Επίση, υπάρχουν πολλέ καπετάνισε πια και αξιωματικοί στα πλοία που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και είναι πολύ καλό λοιπόν να ε, τονίσουμε αυτό το θέμα σε σχέση με την ΕΜΣΑ και για την ισότητα των φύλων και την ισορροπία μεταξύ του. Αυτέ ήταν οι παρατηρήσει μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Κύριο Καραμίτσο. Uh, Μια στιγμή. η κυρία Γιάλα Σέντερ θα πρέπει να πει κάτι προηγουμένως. Παρακαλώ, αν μπορείτε, αν μπορείτε να μου λέτε ότι θέλετε να το λόγο, γιατί στα τηλεπαθητικά δεν τα πάω πολύ καλά. Συγγνώμη, συγγνώμη, ήθελα να, κάνω την, ε, να, να, να δείξω τι είμαι ευγενική και περίμενα να μιλήσουν όλοι οι συντονιστές. Και εγώ. Να συγχαρώ τον συνάδελφο Στάιν για την πρότασή του και για όλη τη δουλειά που έκανε. Να βελτιώσει έναν οργανισμό που Τον προσέχουμε ιδιαίτερα σε αυτήν την Επιτροπή. Διότι εμείς ε, ξεκινήσαμε εξαιτίας όλων των ε, καταστροφών που είχαμε στην Ευρώπη και μετά σιγά σιγά μεγαλώσαμε και αντιμετωπίσαμε τις κρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επαναλαμβάνω αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπιλμπάο για να μπορέσουμε να ε, επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες και στις ε, offshore πλατφόρμες ε, και στις ε, ολικές εγκαταστάσεις που είναι και αυτές offshore που συνεχώς αυξάνονται για να μπορέσουμε να αποφύγουμε προβλήματα ασφάλειας. Αλλά βέβαια για τα κάψιμα τώρα μόνο τις πλατφόρμες έχουμε. Ο εισηγητής εξέτασε με ενδιαφέρον την πρόταση που έκανα για να κάνω έναν παραλληλισμό με αυτό το οποίο συμβαίνει στην αεροπορία όπου έχουμε μια συμβουλευτική επιτροπή. Αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει την έμψα. θα εκτιμηθούν αυτές οι προτάσεις που κάνουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή σχολή κατάρτισης ναυτικών, μια κοινή ακτοφυλακή και πάει λέγοντας. Αυτά είναι καλά για την κοινωνία. Και αυτό το συμβούλιο που εγώ προτείνω, δηλαδή ανοίγει, δίνει προοπτικές για διάλογο στον οργανισμό. Βέβαια οι διάλογοι πολλές φορές ήταν φιλικοί, άλλες φορές λιγότερο φιλικοί. Του εύχομαι, πάρα πολλά, του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Του εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο στο, στους νέους δρόμους που θα ακολουθήσει και τον θυμίζω ότι περάσαμε πολλά από κοινού στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ο κύριος Καραμίτσος. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν ε, κάπως καθυστερήσει τα πράγματα. Τώρα βρισκόμαστε στο επίπεδο προεπιλογής του νέο διευθυντή τη ΕΜΣΑ γιατί ο κύριο Ρόιτερ αποφάσισε να φύγει λίγο νωρίτερα παρά τα θετικά πράγματα που έχει κάνει. Και εμείς από δική μα πλευρά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συγητή και του κοιόδη εισηγητέ για την πολύ καλή δουλειά του και τι καλέ συμβαστικέ τροπολογίε. Δεύτερον, υποστηρίζουμε όλα αυτά τα θέματα που υποστήριξαν σε σχέση με την ε, εκπαίδευση, την αμοιβή αναγνώση πιστοποιητικών, την αντιμετώπιση της πειρατεία κτλ. Έχουμε τώρα κάποιες παρατηρήσεις. Μία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ίσως για σας. Καταρχήν το θέμα που έθιξε, ο κύριος Τέιλορ για τη διάζωση. Για να αναλάβει η ΕΜΣΑ τα θέματα διάσωσης. Αυτό είναι ένα λειτουργικό ζήτημα. Είναι κάτι που κάνουν ήδη ακτοφυλακές σε όλη την Ευρώπη και η ΕΜΣΑ με τους πόρους που έχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επομιστεί αυτό το καθήκον αυτό βέβαια που μπορεί να κάνει η ΕΜΣΑ είναι να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στα κράτη-μέλη όταν εμπλέκονται σε τέτοιες επιχειρήσεις διασώσεως. Το ίδιο ισχύει και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Αυτό είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, πρέπει να προχωρήσουμε βήμα με βήμα και πάλι η ΕΜΣΑ δίνει πολύ καλές πληροφορίες στις ακτοφυλακές των κρατών μέλων της Ευρώπης και στη Μεσόγειο αλλά και στη Βόρεια Θάλασσα για να τις βοηθήσει σε ορισμένα καθήκοντα που μας ενδιαφέρουν. Τώρα το κύριο σημείο για το οποίο έχουμε κάποια ανησυχία είναι οι εγκαταστάσεις εξόριξης οι υπεράκτιες. Γιατί θεωρούμε ότι αυτές οι τροπολογίες που προέρχονται από την Επιτροπή σας μπορεί να ξεφεύγουν από τις τωρινές και στο άμεσο μέλλον δυνατότητες της ΕΜΣΑ και θα υπερφορτώσουν το προσωπικό τους <clears throat> με θέματα όπως πραγματικά τον αξιολογούν τα εθνικά σχέδια αντιμετώπιση εκτάκτων κρίσεων. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ικανότητα προς το παρόν και όπως αναφέραμε και την προηγούμενη φορά χρειαζόμαστε να έχουμε μια πρόταση η οποία θα εξασφαλίσει το ότι θα υπάρχουν ευρωπαϊκές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό και μετά μπορούμε να επιφορτήσουμε την έμψη κάποιον άλλο φορέα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιου είδου ευρωπαϊκού χαρακτήρα αρμοδιότητες και όταν λέμε ότι η ΕΜΣΑ θα πρέπει να συντονίζει τι δράσει των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν τη ρήπανση, αυτό ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει χωρί να υπάρχουν οι απαραίτητε αρμοδιότητε. Αυτό μπορεί να κάνει η ΕΜΣΑ και αυτό γίνεται, είναι αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποιο ατύχημα με ρήπανση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε του πόρου μα για να συντονίσουμε τι αντιρρυπαντικέ αρχέ των κρατών μελών. Εκεί η ΕΜΣΑ σίγουρα μπορεί να βοηθήσει να επιληθεί ένα πρόβλημα. Το θέμα του ανεξάρτητου, της ανεξάρτητας εποπτείας, στο θέμα αυτό θα πρέπει να δούμε εάν και κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει. <clears throat> Αν τώρα ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν την πρωτογενή ευθύνη και στη συνέχεια θέλουμε κάποιον απ' έξω να ελέγχει τα κράτη-μέλη, αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε. από τη στιγμή που η Κομισιόν θα είχε αρμοδιότητα στον τομέα αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε παραδείγματο τα το ατύχημα που έγινε στον κόλπο του Μεξικού και μετά από τι συζητήσει που έγιναν σε αμερικανικό επίπεδο. Εμεί δεν έχουμε μια αντίστοιχη αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω αυτά που έγιναν στι ΗΠΑ. Σας έχουμε λοιπόν πρώτα τι αρμοδιότητε και θα δούμε τι μπορεί να κάνει η ΕΜΣΑ στον επόμενο γύρο αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια ανεξάρτητη εποπτεία πιανού πράγματος όταν δεν έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Αυτό είναι το μόνο σημείο όπου έχουμε κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τις συμβαστικές τροπολογίες. Στα υπόλοιπα σημεία νομίζω ότι μπορούμε να αποδεχθούμε την διατύπωση που, στην οποία έχει φτάσει ο εισηγητής με τους κοιόδους και σας ευχαριστώ τα μάλα. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θα κάνω κατάχρηση της θέσης μου ως ε, Πρόεδρο και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντερόιτερ. Εάν θέλει να πει κάτι. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχάς όλα τα μέλη της Επιτροπής σας που μίλησαν με τόσο καλά λόγια για την ΕΜΣΑ και τον απερχόμενο διευθυντή της. Χαίρομαι που από ό,τι φαίνεται δεν σας απογοητεύσαμε. Οι προτάσεις του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικές. Και χαίρομαι που το θέμα της εκπαίδευσης και της ε, των του ναυτικού επαγγέλματος είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι μάλιστα κατά κάποιο τρόπο ορφανό. Κανείς δεν διεκδικεί την πατρότητά του, αλλά είμαστε στο σημείο να λάβουμε συγκεκριμένε πρωτοβουλίες. Επί του μάλλον πολύπλοκου θέμερος των θαλασσίων εξεδρών έχω μια πρόταση. Στην προφορική τροπολογία Β, στο τέλος της το κείμενο λόγω για συντονισμό της ε, αντιμετώπισης θαλάσσιας ρήπανσης. Ε, ελπίζω στα αγγλικά τουλάχιστον να μην ε, ερμηνευτεί το κείμενο ως συμβολή στη ρήπανση. Εμείς έχουμε 20 πλοία για το σκοπό αυτό, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ρόλος της ΕΜΣΑ είναι να συμβάλλει στον καθαρισμό των πετρελοκυλίδων για παράδειγμα το ποιος θα συντονίσει την επιχείρηση επιτόπου βάσει των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, η εθνική αρμόδια αρχή που, του κράτους που πλήττεται περισσότερο είναι αρμόδια για τον συντονισμό. Οπότε θέτω στην κρίση σας τη σκέψη αυτή. Ότι έμψα δηλαδή θα συμβάλλει ενεργά και αποφασιστικά στον καθαρισμό και θα συντονίσει γενικότερα την ανταπόκριση των κρατών μελών. Και ως Φλέκενστάιν. Α, έχω μια ερώτηση προηγουμένως. Θα ήθελα να βεβαιωθώ ότι ο συνάδελφός μας προς τα εκεί ε, κατάλαβε, κατάλαβε ακριβώς την προφορική τροπολογία που θα υποστηρίξω. Η τροπολογία μου δεν αναφέρεται στην έρευνα, σε δραστηριότητες έρευνας, μόνο διάσωσης. Μόνο διάσωσης. Ε, ελπίζω να διευκρίνησα αυτό που θέλω να πω. Θέλετε Α, δυστυχώς, λέει ο κ. Καραμίσο, κοιτάξτε, στην ε, ιδιολεκτό μα έρευνα και διάσωση πηγαίνουμε, πηγαίνουμε, πηγαίνουμε μαζί. Αυτό που θα στείλει ελικόπτερα για, για την έρευνα θα κάνει και τη διάσωση. Δεν είναι δουλειά τη Έμσα αυτό. Η Εθνική Αρχή του Πρακτικού κράτου Μέλους έχει αυτή την αρμοδιότητα και έχει και τα μέσα στη διάθεσή τη να προβεί σε διάσωση. Η ΕΜΣΑ απλώ έχει τα συστήματα πληροφόρηση μέσω του AIS και άλλων συστημάτων η ΕΜΣΑ ενημερώνει και επικουρεί τα κράτη-μέλη στη διαδικασία αυτή. Αλλά ότι η ΕΜΣΑ, τώρα πει ότι η ΕΜΣΑ έχει αεροπλάνα και ελικόπτερα για έρευνα και διάσωση, όχι. Αυτό δεν είναι δουλειά της ΕΜΣΑ. Τουλάχιστον η ΕΜΣΑ δεν το κάνει ως σήμερα. Τώρα αν ε, η ΕΜΣΑ αποκτήσει εκτοφυλακή στο μέλλον, τι να σου πω, θα δούμε τι οργανισμό θα προκύψει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία, η ώρα του κ. Φλέκενστάιν. Μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Βέβαια δεν περιλαμβάνεται όλα στις ε, συμβιβαστικές λύσεις, αλλά δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε, να υποβαθμίσουμε και αυτά τα οποία συζητάμε, όπως είναι η αντιμετώπιση της πειρατείας, όπως είναι η ασφάλεια στη θάλασσα κτλ, η κατάρτιση η εκμετάλλευση, είπε ο μιλητής στην αρχή, διόρθωση είναι η κατάρτιση. Είναι θέματα τα οποία ακόμα και αν γίνονται μονάχα με προωθούνται με αίτηση των κρατών μελών και της Κομισιόν, πάλι καλά που γίνεται αυτό. Εδώ με ενοχλεί πολύ η συζήτηση που γίνεται δίπλα το πηγαδάκι. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Sorry. ja. Hij stopt er nou mee omdat jullie zitten te praten. Also nogmaals, vielen dank aan die berichters. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδους εισηγητές. Ίσως μπορούμε να συναντιόμαστε η οι, οι άνδρες από την Επιτροπή και να μπορέσουμε να λύσουμε μερικά προβλήματα. Αλλά η κυρία Μπιλμπάου παρόλα αυτά έχει πολύ δίκιο στην παράγραφο 137 θα την ακολουθήσω. Ε, εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Αύριο ψηφίζουμε και θα πάμε στην Ολομέλεια το Νοέμβριο, αν θέλει ο Θεός και αν υπάρξει συμφωνία ο εισηγητής μπορεί ακόμα να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια συμφωνία πρώτης ανάγνωσης με το Συμβούλιο και τότε θα έρθουμε και πάλι στους συντονιστές για την έγκριση. Επόμενο θέμα, η έκθεση Μαρινέσκου για την πολιτική ανταγωνισμού. Είναι μια γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μήπως μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία. Συγγνώμη κύριε Μαρινέσκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Πιστεύω ότι οι περισσότερες τροπολογίες έχουν προστιθέμενη αξία στη γνωμοδότηση. Σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές έχω προτείνει έναν συμβιβασμό ο οποίος έγινε δεκτός. Δηλαδή πέρα από την, δημιουργία του ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου, το, την ε, συγκρότηση αγοράς κτλ. Η τροπολογία αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών, στην εναρμόνιση της παροχής υπηρεσιών και στις κοινωνικές, στα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Για τις αερομεταφορές έχουμε τροπολογίες για τις κρατικές ενισχύσεις, για την δυνατότητα των επιβατών να καταθέτουν, να κάνουν μήνυση και επίσης ε, για το θέμα των αγορών στα αεροδρόμια και την παρακολούθηση των, ενισχύσεων, των κρατικών ενισχύσεων στις low cost αεροπορικές εταιρείες. Για τα δικαιώματα των επιβατών ε, είναι, είναι πολύ σημαντικά στη γνωμοδότησή μας. Αναφέρουμε επίσης την ανάγκη εναρμόνισης του ευρωπαϊκού συστήματος των ε, ξενοδοχή, της στέγασης στον τουρισμό, και μιλήσαμε επίσης για την ανάγκη ο ανταγωνισμός, να αποφύγουμε ο ανταγωνισμός να οδηγήσει σε ένα κοινωνικό ντάμπινγκ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Ευχαριστώ κυρία Μαρινέσκο. Ο κύριος Κεντράου; ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνούμε με την έκθεση Μαρινέσκου αλλά επιτρέψτε μου όμως να εκφράσω την έκπληξή μου ως προς τον συμβιβασμό. Αναγνωρίζω ότι ο εισηγητής κάνει μία απόπειρα αλλά εμείς δεν έχουμε εμπλακεί ποτέ σε αυτή τη στην ε, σύνταξη της ε, συμβιβαστικής τροπολογίας. Θα θέλαμε λοιπόν πριν προχωρήσουμε σε έγκριση τροπολογίας επί του συμβιβασμού τουλάχιστον να μας διαβουλευτείτε για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε την πρότασή μας να προσαρμόσουμε την συμβιβαστική τροπολογία. Η πρώτη συμβιβαστική τροπολογία έχει ένα σωρό ωραία πράγματα. Αλλά στην τροπολογία μου μιλούσαμε για τη σημασία της δημόσιας υπηρεσίας. Δεν το ξαναπαίρνουμε εδώ στο κείμενο. Όταν μιλάμε για ανταγωνισμό και αξιολόγηση, δεν μπορούμε μόνο να μιλάμε για λειτουργία της αγοράς ως τέτοια. Πρέπει να ε, επιμείνουμε ότι θα πρέπει να παρέχονται καλές υπηρεσίες στους χρήστες και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους σιδηροδρόμους, ισχύει για όλες τις ε, μεταφορές. Αυτά ήθελα εγώ να πω, θα ήθελα να προσθέσουμε καινούργια πράγματα σχετικά και να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε καλύτερα, όντας επαφή φυσικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Διμπέκερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ε, εκτιμάμε ιδιαίτερα την δουλειά του κυρίου Μαρινέσκου ως και όδης εισηγητής για την ΑΛΔΕ. Έχω και εγώ καταθέσει τροπολογίες που αφορούν κυρίως στο άνοιγμα της ε, ευρωπαϊκής αγοράς στις διάφορες μεταφορές. Και ο εισηγητής έλαβε υπόψη του τις ε, τροπολογίες. Μιλάμε για τον έλεγχο της ε, ε, άμεσες και έμεσης κρατικές ενισχύσεις οι οποίες αποτελούν φραγμό. Έχουμε επίσης τροπολογίες για τους σιδηροδρόμους. Ο κύριος Τρεμός επίσης συμμετείχε για τις αερομεταφορές. προσπάθησα για λόγους διαφάνειας να προχωρήσουμε ε, στην ε, διάκριση και για το καμποτάζ είμαι απαγοητευμένος. Θα ήθελα να υπάρχει χώρο στο κείμενο και για το καμποτάζ. Τώρα για αυτά που έλεγε ο κύριος Ελχαδράου για το συμβιβασμό. Πράγματι, πρέπει να ξαναδούμε την μεθοδολογία. Για τα υπόλοιπα δεν έχω κανένα πρόβλημα σχετικά με την πρόταση που έχει διατυπωθεί και όπως έχει διατυπωθεί. Περιμένουμε λοιπόν την ψηφοφορία αύριο. Κύριος Κράμερ. Και εγώ θα ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές για τις συμβαστικές ε, λύσεις. Εγώ νομίζω ότι το θέμα της προστασίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να, να εξασφαλιστεί θέματα χάρη όπως η μετακίνηση ατόμων με προβλήματα είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι προϊόν πρόνοιας και να μην κοιτάμε μοναχα τα θέματα του ανταγωνισμού. Κύριε Ρικέ, για την τροπολογία 15 συμφωνούσαμε όλοι ότι οι αρχές ρυθμιστικές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Και τώρα το έχουμε εδώ. Το έχουμε πετύχει και εσείς θέλετε τώρα να το διαγράψετε αυτό. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω την τροπολογία 15. Γιατί θέλετε να μην είναι ανεξάρτητη αρχή. Και ο κύριος ε, Μπαχ βλέπω ότι υποστηρίζει μια φορολογία που επιβαρύνει στη Γαλλία πάρα πολύ με φορολογία τις ξένες επιχειρήσεις και ορισμένες άλλες επιχειρήσεις όπως ο σταθμός του Μιλάνου ε, εφαρμόζουν τέτοιου είδους φόρους. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αρχή των περιφερειακών αεροδρομίων. Μπορεί κανείς να πάει λοιπόν από ένα μικρό αεροδρόμιο σε ένα άλλο αεροδρόμιο. Εμείς μπορούμε να, <clears throat> να λέμε ότι θα, εκδώσουν, θα καλύψουν τόσα εισιτήρια και στην πράξη βλέπουμε ότι ελάχιστα πληρώνονται από τους ίδιους τους καταναλωτές τα περισσότερα είναι επιδοτούμενα από τις αρχές. Προφανώς μπορούν να είναι φθηνότερα αυτά τα αεροδρόμια, αλλά πρέπει να υπάρχουν ορισμένε προδιαγραφές. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλές ε, ε λύσεις για τα θέματα καθυστερήσεων ε, των, τρένων. Για τα αεροπλάνα ξέρουμε ότι μετά από 3-3,5 ώρες υπάρχει αυτή η αποζημίωση. Για του σιδηροδρόμου δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει όμω να έχουμε επομένω μια αρχή η οποία θα εξασφαλίζει ότι όταν υπάρξει μια καθυστέρηση, όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα για ένα ε, καταναλωτή, να μπορεί κάποιο να πάρει το τηλέφωνο, να μιλήσει με κάποιον, να πάρει μια απάντηση, να ξέρει ο καταναλωτη ότι υπάρχει και κάποια αρχή η οποία μπορεί να διαμεσολαβήσει, να παίξει μια ανεξάρτητη διατηρητική λειτουργία και όχι απλω ο κοσμο να, να φωνάζει και να βρίζει. Αυτά. Ε, πρόεδρε, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το είπε ο συνάδελφος Κρέμερ. Λένε ότι βασικά δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο κειμένων. Ελπίζω να με ακούτε. Με ακούτε. Το πιο σημαντικό πάντως για όλους τους, τις μεθόδους μεταφορών είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο κοινωνικός ιστός πρέπει να προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες μας. Πούμε λοιπόν ότι αυτό δεν το έχετε λάβει υπόψη σα. Το κοινωνικό κόστος δεν το έχετε συμπεριλάβει. Συζητήσαμε το πρώτο πακέτο. Τώρα, στην έκθεση αυτή λέτε ότι οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλάβουμε το κοινωνικό κόστος σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, σε όλα τα μεταφορικά μέσα. Μην το ξεχνάτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλει κανείς να απελευθερώσει όλες τις μεταφορές, τον τουρισμό και το κατεξής. Δεν πρέπει λοιπόν να παραβλέψει κανείς το κοινωνικό κόστος. Κύριε Σουρικέ. Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον Μερνέσκου. Πιστεύω ότι αποτυπώνει πολύ καλά την κατάσταση στην αγορά και προς τον Σάλφο Κράμπερ να πω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητούμε τι τροπολογίε. το 1, όχι το 15. Εγώ έχω υποβάλει την υπαριθμόν 5. Εκεί υπογραμμίζω τη σημασία για τις εθνικέ ρυθμιστικέ αρχές να συμβάλλουν στον ευρωπαϊκό συντονισμό. Αυτό είναι προπόθεση πριν την απελευθέρωση. Δηλαδή να ενισχύσουμε το αρχικό κείμενο καταρχήν και να βγάλουμε από τη συζήτηση κείμενα τα οποία είναι λιγότερο απαιτητικά. Η δική μου πάντως είναι η η τροπολογία. Ευχαριστώ. Άλλος. Όχι. Οπότε, κύριε Μπρόνς, από την Κομισιόν. Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο σχόλιο για τις τροπολογίες. Πολύ ωραία. Κύριος Μαρινέσκου. Πρόεδρε, ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Πως τον κύριο Ελκαντράουε να πω ότι η συμβαστική τροπολογία επετεύχθη μετά από διαβούλευση με όλου του συναδέλφους που είχαν υποβάλει τροπολογίες για κάθε εδάφιο ξεχωριστά. Το γραφείο του κ. Ελκαντράουι μας ανακοίνωσε ότι ο κ. Ελκαντράουι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο συμβιβασμό παρά το και ότι αναφέρεται ποιότητα των υπηρεσιών σε σύνδεση με τα κοινωνικά πρότυπα για τους υπαλλήλους κλπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για το ίδιο, το ταυτόσιμο κείμενο, αλλά το τμήμα του κειμένου του συναδέλφου έχει συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά. Πάμε γρήγορα. Αύριο είναι η ψηφορία. Στην Ολομέλεια... Α, μισό λεπτό. 22 Νοεμβρίου στην Επιτροπή θα το θέμα και δεν ξέρω εάν θα προλάβει να πάει στην Ολομέλεια. Κύριε Λίχτεμπερκ ε, είναι καθοδόν, αν δεν κάνω λάθος, οπότε ας διακόψουμε για 10 λεπτά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 So, as you all saw, Όπως είδατε, ήρθε εγκαζομένη κυρία Λίχτεμπεργκ. Εάν λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Τα PNR τώρα, γνωμοδότηση για τα προσωπικά στοιχεία των επιβατών, τα γνωστά ως PNR, κυρία Λιχτεμπέργερ. Να σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε ακόμα ψηφοφορία στην Νομική Επιτροπή και πάντα γίνονται τα θέματα που είμαι υπεύθυνη την ίδια ακριβώ ώρα σε δύο επιτροπές συγχρόνως. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλου αυτού που κατέθεσαν τροπολογίε σε αυτή την ε, γνωμοδότηση 200 τροπολογίε περίπου. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό έχει γίνει αυτό το θέμα και καταδεικνύει απόλυτα το πόσο καυτό και ενδιαφέρον αυτό το θέμα που βρίσκεται στην, ε, <clears throat> ουσιαστικά στη διαδραστική επιφάνεια μεταξύ μεταφορών και καταπολέμησης της τρομοκρατίας αλλά επίσης και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κτλ. Έχουμε συσσωρεύσει αρκετή τεχνογνωσία στα θέματα αυτά, συζητώντας με, με αεροπορικές εταιρείες και με τους υπευθύνους των συστημάτων κράτησης θέσεων στα αεροπλάνα. Δυστυχώς τώρα, εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα να συγκαλέσω μια συνάντηση των συντονιστών, των σχεδόν συγγνώμη, εισηγητών στο Στρασβούργο την προηγούμενη, προηγούμενη εβδομάδα γιατί ήταν και το θέμα των σαρωτών σώματο σώματος που ήταν στην ημερήσια διάταξη ε, τώρα. Όμως μπορούμε να το κάνουμε, είναι όλοι παρόντες ισχυώδεις εισηγητές. Να μπω τώρα σε ορισμένα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Αλλά θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών ώστε το ταχύτερο δυνατό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την ε, επεξεργασία του θέματος αυτού. Η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών επίσης ε, έχει καθυστερήσει για να μας δώσει μια γνωμοδότηση. Έχουμε λοιπόν, διάφορα σημεία τα οποία προέκυψαν από τις προηγούμενες συζητήσεις και θα προσπαθήσω να τα αναφέρω εν συντομία. Το πρώτο ερώτημα είναι πέραν της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να περιλάβουμε και μία ασαφή μάλλον διατύπωση όπως σοβαρή ή βαριά εγκληματικότητα. Επομένως, το ερώτημα είναι μια τέτοια διατύπωση μπορεί να εξασφαλίσει η ασφάλεια δικαίου. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε και για, του, για τα υποκείμενα δικαίου, για τους πολίτες μας και το πώς θα τους αντιμετωπίσει αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό θέλω να έχω την ευκαιρία να συζητήσω με αυτούς οι οποίοι έχουν καταθέσει τροπολογίες, γιατί εκεί που υπάρχει η σοβαρή και η πολύ σοβαρή εγκληματικότητα, τα κράτη-μέλη έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν τι είναι σοβαρή εγκληματικότητα και θα καταλήξουμε σε ένα τεράστιο μπάχαλο ενδεχομένως. Σε κάποια κράτη-μέλη, παραδείγματο χάρη, μια απάτη μπορεί να είναι ένα σοβαρό αδίκημα, αλλά ένας απαταιώνα δεν είναι αυτός που μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων. Αν δω επίσης τη συζήτηση που έχει λάβει η χώρα στο παρελθόν, βλέπω ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε το εξή. ότι δεν είναι μονάχα τα στοιχεία των επιβατών και η επεξεργασία των στοιχείων των επιβατών που μας δίνει τη μόνη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα. Υπάρχει συνεργασία των δικαστικών αρχών, υπάρχουν διαδικασίες συγκεκριμένες που προβλέπονται. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσουν από κοινού <clears throat> και όχι να τα φορτώσουμε όλα στα στοιχεία των επιβατών. Να μην έχουμε λοιπόν την εντύπωση ότι εάν εμείς περιορίσουμε την προσοχή μας στην ε, τρομοκρατική δραστηριότητα και μόνο, θα ανοίξουμε διάπλατα τις πύλες σε άλλες μορφές εγκληματικότητας. Γιατί αυτή η φυσιολογική, αν το μπορώ να το πω έτσι, εγκληματικότητα που εξακολουθεί να υπάρχει, αντιμετωπίζεται με στοιχεία συνεργασίας μεταξύ των διοκτικών αρχών και υπάρχουν επιτυχή μέτρα τα οποία έχουν ε, αντιμετωπίσει αυτή την εγκληματικότητα και δεν εξαρτώνται από τα στοιχεία των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Αυτό είναι μια διευκρίνηση λοιπόν που ήθελα να κάνω. Επίσης πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εισαγωγή μιας νέας μορφής ορισμού για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αρχικές διατυπώσεις που είχαμε στο παρελθόν για να μην δημιουργήσουμε πολυπικιλία ερμηνεών στα κράτη-μέλη και υποσκάψουμε την ασφαλεία δικαίου για τα θέματα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σημείο το οποίο είναι σημαντικό για μένα. Αλλά σας είπα και πάλι ότι θα ήθελα να προσπαθήσω να συζητήσω με αυτούς που κατέστησαν τις τροπολογίες και να καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική λύση. Ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το ερώτημα push and pull, όθηση ή έλξη. Εδώ υπάρχουν δύο τάσεις. Εμείς στην Ευρώπη θέλουμε να υπάρξει η προώθηση των στοιχείων, στο, το αντίστοιχο η έλξη των στοιχείων δεν πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ότι κάποιος δηλαδή έχει το δικαίωμα μόνος του να πάρει τα στοιχεία από το σύστημα κράτησης ε, θέσεων επιβατών. Κάτι το οποίο είναι ακόμα ξένο με την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση για το δίκαιο, ενώ στις ΗΠΑ είναι διαφορετικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι <clears throat> κάποιες αεροπορικές ε, εταιρείες δεν μπορούν ακόμα να εξασφαλίσουν κάτι τέτοιο και γι' αυτό θα πρέπει να αναμείνουμε λιγάκι. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στην αντιμετώπιση μας για να μην δημιουργήσουμε διαφορετικά πρότυπα νομικά μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τίθεται το ερώτημα του τι γίνεται με μια αεροπορική εταιρεία που δεν παραδίδει τα απαραίτητα στοιχεία. Ο κύριος Ρικέ είχε καταθέσει μια ενδιαφέρουσα τροπολογία που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, κάποιες προσωρινές κυρώσεις, αλλά αυτό να μην σημάνει ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια της εταιρεία αν για κάποιο τεχνικό λόγο δεν μπορούσε να δώσει αυτά τα στοιχεία. Και αυτά είναι σημεία τα οποία τα έχουν θίξει πολλοί από τους καταθέτες των τροπολογιών. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ομάδα από τροπολογίες οι οποίες ασχολούνται με το θέμα του παρατήματος και των στοιχείων που θα πρέπει να παραμείνουν οριστικά μέσα στο παράτημα. Και εδώ θα ήθελα κυρίως να συζητήσω με τους δύο κύριους καταθέτες τροπολογιών για το παράτημα και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή συμβιβαστική τροπολογία η οποία θα μας ε, βοηθήσει να αποτρέψουμε να κάνουμε 80 ή κάτι τέτοιο με μονομένε ψηφοφορίες. Και φαντάζομαι ότι και αυτοί που κατέστησαν τροπολογίες θα αναφέρουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω. Περιμένω καλύτερα να ακούσω τις προτάσεις σας και τις ερωτήσεις και όπως σας είπα θέλω να κάνουμε μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και δεύτερον να μιλήσω και με τους ε, καταθέτες τροπολογιών, είτε βρίσκονται στην Επιτροπή μας, είτε είναι εκτός αυτής, για να καθορίσουμε τις λεπτομέρειες των συμβαστικών. δε Grandes Pascual. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις οικουμενικές αξίες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και έχει ως θεμέλιο την αρχή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η τρομοκρατία αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις όλων αυτών των χαρκών. Το τα στοιχεία PNR μπορούν να χρησιμεύσουν για να καταπολεμήσουμε ουσιαστικά αυτά τα διεθνή εγκλήματα. Προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο σύστημα ελέγχου των επιβατών με το ΑΠΗ, με τα συστήματα USS VHS και είναι πολύ πιο αξιόπιστα τα στοιχεία PNR από ότι τα στοιχεία API. Εμείς σε αυτήν την Επιτροπή καυγαδίζουμε για θέματα ουσίας ε, τα οποία είναι, ναι, σωστό, είναι σωστό να γίνεται αλλά εμάς δεν είναι αρμοδιότητά μας αυτή η έκθεση είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Τώρα για τις ε, καθαρά ε, περιορισμένες αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής μας θα έχουμε λίγες δυσκολίες με την εισηγήτρια. Η κυρία Λίχτεμπερκ περιορίζει το εφαρμοστικό πεδίο τόσο ώστε την ε, τροποποιεί και την απογυμνώνει από όλε τι τις αξίες που θα ήταν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Δεν συμφωνώ με τις τροπολογίες της. μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Κατά τα άλλα, η συγγήτρια κράτησε, αυτά, κράτησε τα στοιχεία έλαβε συγγνώμη υπόψη της το άρθρο 29 και τα βασικά στοιχεία για την προστασία των ανθρωπίν των ε, ε, προσωπικών πληροφοριών. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τους υπόλοιπους συναδέλφους της ομάδας για, τις, για τα άρθρα της οδηγίας. Μπορούμε να έχουμε περιθώριο λάθους. Θα έλεγα ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πρέπει να συμπληρώνουν περισσότερα στοιχεία από αυτά που λαμβάνουν μέχρι τώρα από τους επιβάτες μέσω των διαφόρων συστημάτων συλλογής πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να έχουμε δυσαναλογία. Θα μπορούσαμε για λόγω του όγκου της μεταφοράς ε, ε, δεδομένων να μην έχουμε τις, ε, τις πτήσεις Ε, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία των ανταποκρίσεων. Εγώ στην, ως μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών θα κάνω πολύ περισσότερες τροπολογίες από αυτές τις οποίες θα κάνω εδώ. Εγώ θα έλεγα στην εισηγήτρια να συνεδριάσουμε για αυτό ε, το θέμα αλλά και για άλλα και γι' αυτό βέβαια που δεν συναντηθήκαμε δεν έφταιγε η συγγήτρια ούτε κανένας άλλος απλώς ε, ο φόρτος εργασίας του Κοινοβουλίου. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε τι, ως Επιτροπή Ουσίας μπορούμε να αναλάβουμε τέτοιο πράγμα. Κανένας δεν μπορεί να στερήσει από τον άλλον τη δυνατότητα γνωμοδότησης και τροποποίησης αν καταλήξουμε σε συμφωνία, κυρία εισηγήτρια, εμείς θέλουμε να σας κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πολύ κοντά. Κυρίως ε, για τις ε, προτάσεις σας εκείνες που αφορούν στην Επιτροπή Μεταφορών. Και μετά, για τα υπόλοιπα, θα πρέπει να αποφασίσουμε να συζητήσουμε εφόλης της ύλη ή να περιοριστούμε μόνο στα θέματα που αφορούν στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Τικάου. Υποστηρίζω απόλυτα την κυρία Λίχτεμπέργκερ. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό ο οποίος να συσπυρώσει μεγάλη πλειοψηφία. Εγώ κατέθεσα πολλές τροπολογίες που ζητούσαν η ανάλυση των στοιχείων PNR να χρησιμεύσουν μόνο για την διαπίστωση των τρομοκρατικών πράξεων και στις έρευνες. Εγώ ζήτησα η διαβίβαση στοιχείων να περιοριστεί μόνο στη χρήση τους για να διαπιστώσουν συγκεκριμένα τρομοκρατικές πράξεις κατά την ανακριτική διαδικασία και στα δικαστήρια. Θα ήθελα η κράτηση των στοιχείων να είναι περιορισμένη μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών για να σεβαστούμε και την οδηγία που αφορά στις ε, τηλεπικοινωνίες. στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. Επίσης κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι εδώ υπάρχει αντισυνταγματικότητα. Θα συμφωνούσα λοιπόν με την τροπολογία που περιορίζει ακόμη περισσότερο την δυνατότητα κράτησης των στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι απόλυτα μυστικά και οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να διορθώνουν και να σβήνουν τα στοιχεία που τους αφορούν. Και πιστεύω ότι όλες οι διατάξεις που αφορούν στις προσφυγές στα δικαιώματα αποζημίωσης πρέπει να υποστηριχθούν. οι συνάδελφοι γράντε και η κυρία Πέτρα Κάμερ λένε ότι θα έπρεπε να διαβιβάζονται μόνο συγκεκριμένα στοιχεία. Βέβαια υπάρχουν κράτη τα οποία λένε ότι μόνο το 30% των στοιχείων μπορεί να συλλεχθεί και αυτό σε τέσσερα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αναλάβουμε τέτοιου είδους υποχρεώσεις και πρέπει να τις συζητήσουμε. Τα στοιχεία PNR δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς λόγους και χρειαζόμαστε πολύ αυστηρούς κανόνες ασφάλειας για τα στοιχεία PNR. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε την ε, διαβίβαση των στοιχείων PNR προς άλλες χώρες τα στοιχεία πρέπει να αναλύονται μόνο στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια για να γίνεται σεβαστός και ο σχετικός νόμος για την προστασία των, των προσωπικών στοιχείων. Αν αυτά τα στοιχεία έπρεπε να τα διαβάσουμε σε τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουμε μια σαφέστατη ε, συμφωνία με τις ε, συνυπογράφουσες χώρες. Εγώ υποστηρίζω να διαγράψουμε το άρθρο 4 παράγραφος 2 Η οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις. Είμαστε υπέρ της ασφάλειας των επιβατών, είμαστε υπέρ της εφαρμογής αυτών των διατάξεων για να μπορέσουμε να κατεπολεμήσουμε συγκεκριμένα εγκλήματα όπως η τρομοκρατία. Δεν μπορούμε όμως να αποδοπατήσουμε και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων επιβατών. Κύριε Ευχαριστώ πολύ. Και... Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ε, σε μένα είπατε, ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λιχτανμπέργια, την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι πήγε έξοχα. Μου άρεσε το ύφο του κειμένου. Κοιτάξτε, εμείς όλοι εδώ είμαστε σαφώ κατά της τρομοκρατίας. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανεί με την ανάγκη να αγωνιστούμε κατά της τρομοκρατίας. Όμως, τα μέτρα που λαμβάνουμε εδώ και 10 χρόνια ήταν λάθασμένα εν πολύ. Πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Μετά από την 11η Σεπτεμβρίου επικράτησε ε, ένα είδος πανικού όχι μόνο στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και εδώ και εγώ είμαι υπέρ όλων αυτών των μέτρων, έτσι. Δεν υπάρχει εμφαλή περί αυτού. Όμως, κάποιες προτάσεις και κάποια νομοθετικά μέτρα ε, εμπνεύστηκαν μάλλον από πανικό παρά από οτιδήποτε άλλο. Οπότε Γενικώ, ναι, σύμφωνα με το ύφο του κειμένου. Έχω όμω και τι επιφυλάξει μου. Κάποιε γενικέ που αφορούν την ομάδα μου, ε, του φιλελευθέρου, και κάποιε πιο εθνικιστικού αν θέλετε χαρακτήρα, όσο και αν είναι κακιά η λέξη. Μου επιτρέπετε? Μου επιτρέπετε, ευχαριστώ πολύ. Το Λονδίνο μου έδωσε το πράσινο Φώ Λοιπόν, ο κατάλογο ε, εγκληματιών. Ε, καταλαβαίνω τα επιχειρηματά σα. όμως, εάν διαγράψουμε εκεί τα πάντα, θα λέω ότι πιθανότατα αποδυναμώνουμε εντελώς το μέτρο. Στη χώρα μου έχουμε μάθει ότι το διεθνές σοβαρό έγκλημα και η τρομοκρατία πρέπει να συμπεριληφθούν. Διότι, για παράδειγμα, το εμπορίο ναρκωτικών. για να το πω πιο συγκεκριμένα. Εκτός από την τρομοκρατία, έτσι. Ε, πρέπει να συμπεριληφθεί. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν μια συμβιβαστική λύση προκειμένου. Και, και, δεν ξέρω αν το είπε, δεν θυμάμαι αν το είπε η κυρία Λίθενμπεργκερ, αλλά είναι ζωτική σημασία να πούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί σημαντικότατη βελτίωση σε σύγκριση με την περασμένη. Το κείμενο αυτό εδώ είναι πολύ περισσότερο συνεπές και συνεκτικό και πιστεύω ότι το πιστεύουν αυτό και οι περισσότεροι εδώ. Λοιπόν, μετά οι προθεσμίες, οι χρονικέ προθεσμίες ε, διατήρηση των δεδομένων. Πραγματικά ε, δεν ξέρω τι να πω. Ακούστηκαν ένα σωρό διαφορετικές ελλακτικέ λύσεις. Θα δούμε αν προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα συμβαστική λύση. Εγώ θα μπορούσα για τους σκοπούς της ε, γνωμοδότησης ε, να αφήσουμε την Επιτροπή Λίμπε να προκρίνει κάτι. Δεν, δεν έχω πραγματικά άποψη. Είμαι φιλελεύθερος. <laughs> Πάντως κάπου στη μέση πρέπει να βρεθώ τελικά. Τώρα το push pull η λύση Όπω όπως ονομάζουμε, πρέπει να προκριθεί, πιστεύω. Αλλιώ δεν υπάρχει συνέπεια στο κείμενο. Και σίγουρα θα υπάρξουν διαρροές δεδομένων. Και αυτό ακριβώ είναι που δεν θέλουμε. Τώρα, PNR στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες ήθελαν αυτό να αφορά τους πάντες και τα πάντα. Χαίρομαι που αυτό αφορά μόνο την Ευρώπη, Όμω θα έλεγα επιπλέον ότι οι ενταποκρίσεις και οι διελεύσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν. Θα είναι πολύ παράξενο να συμπεριλάβουμε και αυτού του είδους τα στοιχεία. Οπότε προτείνω να το περιορίσουμε στην Ευρώπη. Αυτά είναι και οι βασικές μας ανησυχίες. Έχουμε φυσικά υποβάλει τροπολογίες, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και ω προ τα παραρτήματα. Θα μπορούσα να δεχθώ ότι κάποια από τα παραδείγματα που προαναφέρετε θα μπορούσαν να βγουν σύμφωνοι για ορισμένα, όχι όμως για όλα. Πιστεύω ότι κάποιες εξαιρέσεις δεν είναι σωστές. Έκατα ε, κλείδι, κύριε Πρόεδρε. Το ύφος του κειμένου, όπως είπα, Χρειάστηκαν δέκα χρόνια να καταλήξουμε σε ένα κείμενο. Το ύφο του είναι το σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπράτπο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, θέλω να πω ότι γενικά συμφωνώ με την κατεύθυνση της γνωμοδότησης της κυρίας Λίχτεμπεργκ. Πολλά θέματα συνδέονται άμεσα με την γνωμοδότηση αλλά θα ήταν χρήσιμο να αναφερθείτε και σε μερικά πιο γενικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να πούμε ότι οποιοδήποτε σύστημα PNR θα πρέπει να είναι τμήμα μια πανοπλία που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τι τρομοκρατίες. Έχουμε δεδομένα για τους ε, τρομοκράτες, έχουμε πολύ καλές υπηρεσίες πληροφοριών. Έχουμε μέσα λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Τώρα για τις ιδιαιτερότητε του προγράμματο PNR, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό και έχω παρακολουθήσει και στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών όλα αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι υπάρχουν τρει ιδιαίτεροι τομεί στου οποίου θέλω να εστιάσω την προσοχή μου, ιδίω σε σχέση με τι τροπολογίε. Πρώτα απ' όλα, ξέρουμε όλοι τι θα πει η τρομοκρατία σε γενικού όρου, αλλά τι είναι το σοβαρό έγκλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, να βρούμε ένα σωστό ορισμό όταν εγκρίνουμε κάποια συμβαστική λύση, δεν θέλω να επαναλάβουμε το ίδιο σφάλμα που κάναμε όταν εισαγάγαμε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο υποτίθεται να είναι για τα πιο σοβαρά εγκλήματα και έφτασε να χρησιμοποιείται και για τους λαθρεμπόρους τσιγάρων, παραδείγματος χάρη τέτοιων πραγμάτων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το στόχο που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια να περιορίσουμε την εμβέλεια αυτή της λύση είναι το θέμα της διάδοσης σε τρίτες χώρες. Ανέφερε ο προηγούμενο ομιλητή ότι μιλούσαμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα PNR αλλά δεν μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα και χωρισμένα από άλλες συμφωνίες που έχουμε συνάψει με άλλες χώρες. Αυτό που με ανησυχεί είναι το θέμα του ποιος μπορεί να έχει τη διάδοση αυτών των στοιχείων και κάτω από ποιε μορφές περιορισμών και πώς αντιμετωπίζετε το να εξασφαλίσετε ότι οι φορείς που έχουν αυτά τα στοιχεία δεν θα τα μεταδώσουν σε άλλους, σε τρίτους. Στις ΗΠΑ όταν μιλούσαμε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Είχαν πει ορισμένοι μπορεί να το πάρει και η εφορία αυτό το σύνορο δεδομένο. Μα όχι, δεν είναι τέτοιο θέμα. Αυτά τα στοιχεία για τον αγώνα κατά τη τρομοκρατία. Και πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για τα θέματα αυτά. Για τα θέματα προστασία δεδομένων. Υπάρχει και εδώ χώρο συζήτηση, όπω είπε η κυρία Λίχτεμπεργκ, ιδίω για το χρόνο φύλαξη των δεδομένων αυτών. Υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει γι' αυτό, αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι είναι, όπως λένε και οι δύο φράσεις που έχουμε στις τροπολογίες, υπάρχει μια φάση που λέει να κάνουμε ανώνυμα τα δεδομένα και η άλλη λέει να τα αποεξατομικεύσουμε, να τα αποατομικεύσουμε. Μπορεί να σημαίνει το ίδιο πράγμα, αλλά πρέπει να έχουμε μια ενιαία ορολογία στα θέματα αυτά και εδώ χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, όπως και το θέμα του push and pull. Είναι φανερό, όπως είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιο μέτρο χωριστά από οποιοσδήποτε άλλες συμφωνίες έχουμε. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτό συναρμόζεται με τις άλλες συμφωνίες που έχουν ήδη συναυθεί ή είναι υπό εξέταση για να συναυθούν. Και αν ε, πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Καναδά, αντιμετώπισα πάρα πολύ τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Φαίνεται ότι έχουμε ένα θετικό ιστορικό εκεί και μπορούμε να κοιτάξουμε αυτές τις συμφωνίες, να δούμε αν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πιο επίμαχο θέμα φυσικά είναι το παράτημα. Όπως και οι περισσότεροι, εγώ έχω κάποιες ανησυχίες για τον αριθμό των στοιχείων, τον αριθμό των ε, τετραγωνιδίων που πρέπει να γεμίσει κανείς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα, πιστεύω, Θέλω να σταθώ όμως μονάχα σε μία περιοχή όπου μπορούν να προκύψει κάποια, μπορεί να έχει προκύψει κάποια σύγχυση και χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση. Ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο PNR είναι πληροφορίες για τακτικούς επιβάτες αεροπορικών εταιριών, frequent flyers. Δεν νομίζω ότι αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό. Είναι πιο χρήσιμο να ξέρει κανείς ποιοι είναι οι τακτικοί προορισμοί στους οποίους μπορεί να πηγαίνει κάποιος. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε λοιπόν. Γιατί έχει νόημα να ξέρουμε πού πηγαίνει κάποιος σε τακτική βάση και επομένω αν έλκεται κάποια ε, υποψία από αυτό. Αλλά το αν πετάει κανείς πάρα πολύ συχνά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αν η κυρία Λίχτεμπερκ είναι στο πρόγραμμα ε, τακτικών επιβατών της Λουφτχάνσα της Όστρια, δεν σημαίνει αυτό τίποτα, απλώ σημαίνει ότι πρέπει να έρθει στι Βρυξέλλε κάθε τρει και μία. Αλλά δεν την κάνει αυτό, τρομοκράτησα. Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Ότι χρειαζόμαστε καλύτερου και πιο στεγανού ορισμού στα θέματα αυτά. Και αυτό είναι το έργο στο οποίο πρέπει να προχωρήσουμε πρωτού πάρουμε μια τελική απόφαση για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί ομιλητέ ακόμα, ο κ. Κόλιτσεκ. Πιστεύω ότι όλοι οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλέον υποπτή τρομοκρατίας, διότι ταξιδεύουν συχνά προς τακτικού προορισμούς. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε, πιστεύω ότι από τη μια μεριά έχουμε τις ε, πολιτικές ελευθερίε και από την άλλη μεριά την προστασία από τους τρομοκράτες. Αυτό είναι το μόνιμο θέμα που επανέρχεται στη συζήτηση. Το ερώτημα το οποίο εγώ όμως θέτω τακτικά είναι γιατί δεν ασχολούμαστε με τους βιβάτες στο μετρό για παράδειγμα που ο κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης είναι πολύ πιο υψηλός. Και μετά έχουμε και το θέμα της προστασίας των δεδομένων γιατί σε κάθε χώρα υπάρχουν τέτοιες αρμόδιες ε, αρχές και αυτές οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν νομίζω ότι θα χαρούν αν ε, δουν ότι υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα διαρροή δεδομένων. Εγώ συμφωνώ με την συνάδελφο Τικάου και με τις τροπολογίες που προέτεινε. Αποτελούν μια ιδανική ισορροπία, θα έλεγα. Να πω επίσης ότι η κυρία Λίχτεμπέγκερ όντως έκανε εξαιρετική δουλειά. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η τελική συμβαστική λύση δεν θα χαρακτηρίζεται από υψηλή αποτελεσματικότητα, αλλά τουλάχιστον θα είναι μια καλή λύση. Και Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Λιχτενμπέργκερ. Ε, έχω τις παρατηρήσεις. Πρώτον, πολλές από τις τροπολογίες, κυρίως της εισηγήτριας, αποσκοπούν στην συμπερίληψη της τρομοκρατίας και της μη συμπεριλήψεις του εγκλήματος. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον διάκριση μεταξύ αυτών των δύο. Οι τρομοκράτε χρησιμοποιούν το έγκλημα για να αποκτήσουν οικονομικά μέσα. Υπάρχει μια επικάλυψη, μια μηδέα επικάλυψη και εγώ υποστηρίζω ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Πολλέ φορέ αυτά τα δύο ταυτίζονται. Μπορεί να υπάρχει διάκριση, ανάγκη διάκριση των δεδομένων, σύμφωνοι, αλλά είμαι μάλλον υπέρ της αποτελεσματικότητας πλευράς ασφαλείας. Οπότε να συμπεριληφθεί και το έγκλημα. Για το push pull πιστεύω ότι αυτό δεν επηρεάζει εν τέλει την ασφάλεια των δεδομένων. Έχουμε έναν ε, πομπό, έναν δέκτη, όλα αυτά είναι κρυπτογραφημένα. Δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη και ποιο είναι το κόστος. Όποιοι είναι υπέρ του push, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού, είμαι υπέρ του pull, έχετε την ευθύνη της μεταβίβασης των δεδομένων και του μέσου, το οποίο δεν είναι ο σκοπός αυτής της ιστορίας. Αν οι εταιρείε, οι αεροπορικέ εταιρείε είναι υπέρ του PULL, του push με συγχωρείτε, αυτό δεν μπορούμε να του το επιβάλλουμε. Από την άλλη μεριά, το κόστος και για το push και για το pull, ένα κόστος το οποίο φυσικά κατανέμεται. Το push πάντως δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να επιβληθεί στις αεροπορικές εταιρείε για λόγους ευθύνης αλλά και κόστους. Άλλωστε νομίζω το είπαν και άλλοι. Τώρα, οι τρίτες χώρες και οι απλές ανταποκρίσεις δεν μπορούν να συμπεριληφθούν γιατί το σύστημα αυτό θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο εν τέλει. Και τέλος μια λέξη για τις υπερβολικές κυρώσεις. Να κατάσχει κανείς τώρα αεροσκάφη ή άδειες ε, λειτουργίες αεροπορικών εταιριών ε, είναι απόλυτα υπερβολικό. Υπάρχουν τα άνομα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και αυτό είναι η λύση προκειμένου. Τέλος, το θέμα είναι να πετύχουμε μια συμβαστική λύση εν ώψη της ε, ψηφοφορίας. Το θέμα είναι να καθίσουμε, να δουλέψουμε και να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες. Ας, κάνουμε, ας δουλέψουμε με τους ε, σκιώδεις, ας το συζητήσουν και εσωτερικά οι ομάδες. Αλλά κάτι να κάνουμε, γιατί ο χρόνος πιέζει. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε είπανε ότι είχαμε 219 τροπολογίες ενώ πρόκειται απλά και μόνο για μία γνωμοδότηση. Αυτό αποδεικνύει ότι τελικά το θέμα ανησυχεί ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. Η ΛΥΜΠΕ είχε ζητήσει να αφήσουμε στην ΛΥΜΠΕ όλα όσα αφορούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πράγματι, για τα δυστυχήματα χρειάστηκε να αναρωτηθούμε κατά πόσο οι μεταφορές συνδέονται με την πρόληψη των ατυχημάτων του. Και εδώ πάλι αφορά στις αεροπορικές εταιρείε και στα δικαιώματα των επιβατών. Αυτά τα στοιχεία πιενέρω. Ο κύριος Δεπασκουάλη είπε ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις μεταφορές και σε ό,τι φύγει άμεσα τις μεταφορές και τον τρόπο ταξιδίου. Όλοι λοιπόν συμφωνούμε, το είπε και η κυρία Λίχτεμπεργκ. Κανένας δεν θα χρειαστεί να ζητήσει κάτι το επιπλέον όσον αφορά Τώρα τα στοιχεία και την κράτησή τους, ε, τα σκάνερ ήταν πολύ πιο απλό πράγμα γιατί δεν ε, κατέγραφαν, ε, δεν ε, διατηρούσαν τα στοιχεία. Μιλήσαμε στην τροπολογία 85 γίνεται αναφορά στις ε, βαριές εγκληματικές ενέργειες, εκρηκτικά σωματεμπορία κτλ. Δύσκολα όμως μπορούμε να κάνουμε εμεί διάκριση μεταξύ της διεθνούς τρομοκρατίας και του μεγάλου οργανωμένου εγκλήματος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ο κύριος, Πάρκ, ο κύριος Πίρκελ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο θετικά πράγματα. Και μετά δύο κριτικές. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνε οι αεροπορικές εταιρείες για τη διαβίβαση των δεδομένων δεδομένου ότι οι ταξιδιώτες, οι επιβάτες είναι αυτοί που τα δίνουν στις εταιρείες. Τώρα για τις τρίτες χώρες ε, θα πρέπει να σεβαστούμε κριτήρια ασφάλειας. Χρειάζονται ισοδύναμα επίπεδα προστασίας στα κράτη-μέλη και μόνο σε αυτή την περίπτωση, μόνο αν υπάρχει ισοδυναμία μπορούμε να διαβιβάζουμε στοιχεία. Αυτό που μου φαίνεται πιο προβληματικό είναι το εξής και οι συνάδελφοι μίλησαν γι' αυτό. Δεν μπορούμε εμείς, ε, δεν είναι εύκολο να περιορίσουμε τις δραστηριότητες αυτού του μέσου. Αλλά εδώ το σπάμε στα δύο. Πρόκειται για ένα μέσο που θέλουμε να έχουμε για να εγγυθούμε την προστασία του πολίτη. αποκλείουμε, δεν μπορούμε εμείς να αποκλείσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Άμα αποκλείσουμε το οργανωμένο <clears throat> έγκλημα δεν θα μας χρειάζεται πλέον τίποτα. Θα μπορούσαμε πραγματικά να το ξεχάσουμε ένα τέτοιο κείμενο. Ξέρουμε όλοι ότι... Υπάρχει ρευστή διέλευση από το οργανωμένο έγκλημα με την τρομοκρατία. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε. Είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να επικρίνω είναι το γεγονός ότι εδώ προτείνονται κάποιες προθεσμίες για το, το περιορισμό της κράτησης των δεδομένων που είναι πραγματικά μη ρεαλιστική περιορισμή όταν θέλει κανείς να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα. Αν δεν έχει νόημα λοιπόν να μαζέψει κανείς δεδομένα τα οποία μετά από 30 μέρες τα ξαναπετάει κανείς, γιατί δεν προφταίνει να κάνει τις αναλύσεις που θέλει να κάνει κανείς. Αν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τρομοκρατικές ενέργειες οι οποίες αναπτύσσονται μέσα σε μεγάλα χρονικά διάστημα, 30 μέρες για να κρατήσουμε τα δεδομένα, ουσιαστικά κάνουν τελείως άχρηστη αυτή την οδηγία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητές τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι προθεσμίες κράτησης φύλαξης των ε, δεδομένων πρέπει να είναι μακρύτερη, αλλά φυσικά να λάβει κανείς υπόψη και την καλύτερη προστασία των δεδομένων. Αλλά ο χρόνος φύλαξης πρέπει να είναι λογικός. Κύριε Φώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λίχτεμπεργκερ, που έχασα τη, τη μισή σας παρέμβαση σήμερα το απόγευμα. Απλώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο εξαίρετος συνάδελφός μου, ο κύριος Bradburn. Δεν θα μπρω σε όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν όμως δύο ή τρεις τομείς που αναφέρθηκαν και από άλλους συναδέλφους που χρειάζονται περισσότερη σκέψη από όλους μας για τις τροπολογίες. Το ουσιαστικό θέμα είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. και αν γίνεται σωστά η αντιτρομοκρατική ενέργεια, είναι πολύ λίγα πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνουμε εμείς με την ομοθεσία μας. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω το ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στις υπηρεσίες του Ηνωμένου που ασχολούνται με το θέμα αυτό και είχε έρθει η Σόβι Ιντβέλτ, η οποία ασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα δημοσίων ελευθεριών και συναντήσαμε πολλού υψηλού επίπεδου αξιωματούχους σε αυτούς τους τομείς. Και με ενδιέφερε πάρα πολύ η προστασία των δεδομένων και το πώς εξασφαλίζα την προστασία των δεδομένων και αυτά. Είναι, ήταν λίγες περιπτώσεις που έπρεπε να υπάρξει περαιτέρω εξέταση ενός φακέλου και ήταν πολύ λίγος ο αριθμός των ανθρώπων που είχαν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Πρέπει όμως να υποστηρίξω αυτό που είπε και ο κύριος Πίρκλ για τον χρόνο κράτησης των δεδομένων. Είναι μεγάλο πρόβλημα το να έχουμε μια συγκεκριμένη προθεσμία για τη φύλαξη των στοιχείων αυτών. Γιατί είπανε, φυσικά, η κύρια αιτία που κρατάμε όλα αυτά τα δεδομένα είναι για την τρομοκρατία. Αλλά δεν μπορείτε να ξεχάσετε το θέμα του σοβαρού εγκλήματος, των μεγάλων αθρεμπορίων και όλων αυτών των προβλημάτων που θέλουμε να ξεφορτωθούμε. Πολλές φορές θέλανε 5 ή 6 χρόνια για να μαζέψει κανείς αρκετά στοιχεία για να στείλει κάποιος στο δικαστήριο και μετά στη φυλακή. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω ποιο είναι το σωστό χρονικό πλαίσιο για να κρατήσουμε τα δεδομένα. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικά. Τόσο κοστίζει να μαζέψουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Και στη συνέχεια, το ερώτημα είναι, εμπιστευόμαστε τους φύλακες τις ε, υπηρεσίες των κρατών μας μελών για το αν θέλουν να κρατήσουν τα στοιχεία αυτά περισσότερο όταν χρειάζεται. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια μεγαλύτερη ευκαμψία. Δεν πρέπει να είμαστε ε, να, κάνουμε εκτόσεις παρά το γεγονός ότι είναι, είμαι σύμφωνος ότι πρέπει να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Εν γέννη λοιπόν. για τους ε, τακτικούς επιβάτες. Μας ενδιαφέρει ο τακτικός προορισμός. Αν πηγαίνει κάποιος συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Αν πηγαίνει σε κάποιο μέρος το οποίο είναι επίμαχο. Και πάλι πρέπει να υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη. Αυτοί οι οποίοι εξασφαλίζουν τα συμφέροντά μας, να τους εμπιστευόμαστε ότι το κάνουν στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα σημεία που έχουν τονιστεί. Υπάρχουν μερικοί ακόμα τομεί που δεν είναι σαφείς δεν θα ψηφίσουμε όμω αύριο και θα προλάβουμε ίσω να ξεμπλέξουμε ορισμένα θέματα για να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση. Ευχαριστώ. Το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο. Ο κύριος έχει το λόγο. Πρόεδρε, συγχαρητήρια και από μένα στην εισηγήτρια για ένα κείμενο εξαιρετικά χρήσιμο για τη συζήτηση. Ε, αλλά συγχαρητήρια και για τα θέματα τα οποία πρέπει βεβαίω να συζητήσουμε προσεκτικά. Πολύ έχουμε τις ε, πολιτικές ελευθερίες, αλλά δεν ξεχνούμε κιόλα. Πριν από ένα μήνα ήταν η δέκατη επέτειος της 11 Σεπτεμβρίου. Και α μην ξεχνούμε την 7η Ιουλίου του 2005 στο Λονδίνο, 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκεί. Ή τη Μαδρίτη, 181 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του 11 Μαρτίου του 2004, λίγε μέρε πριν από τις βουλευτικέ εκλογές στην Ισπανία. Όταν λοιπόν κάποιοι μα λένε για πανικό, η αλήθεια είναι ότι είμαστε μόλις ένα βήμα πριν την επόμενη τέτοια καταστροφή. Φυσικά και υπάρχουν πολιτικές για την προστασία των δεδομένων και καλό είναι αυτό, αλλά ε, θέλω κάποιο να μου πει πού γίνεται κατάχρηση, αν υπάρχει στα σημερινά συστήματα. Γίνεται κατάχρηση των σημερινών δεδομένων, των δεδομένων που συλλέγονται αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για φόβο και μόνο ότι θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει ούτε ένα στοιχείο που να μα λέει ότι γίνεται κατάχρηση. Α συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με φανατικού. Με ανθρώπου που δεν διακρίνουν το καλό από το κακό. Ε, μιλάμε για ανθρώπου οι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για να κάνουν το κακό. Αυτή η απειλή είναι εδώ. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα θα είναι αυστηρά. Στη χώρα μου ζήσαμε 30 χρόνια επιθέσεων με τη μορφή βομβών, παγιδευμένων αυτοκινήτων, με τεράστια πόλια θυμάτων. Η απειλή όμως είναι ακόμα χειρότερη σήμερα. Ξέρω ότι υπάρχουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε την τρομοκρατία στην Ευρώπη, αν χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση κλπ. Όχι, ο κόσμος είναι ένας, ενιαίος. Μιλάμε για αεροπορία, μιλάμε για αεροπορικές μεταφορές. Μιλάμε για τρόπους μεταφοράς που δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Άρα ό,τι είναι να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε σε συνεργασία με τρίτες χώρες όπως οι Μέρες Πολιτείες που τηρούν δεδομένα για 50 χρόνια. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω τον κύριο Ρικέ. Τώρα συμφωνώ με τον κύριο Πρίκα. Μαζεύουμε που μαζεύουμε τα δεδομένα με πολύ ψηλό κόστος. Γιατί να με χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση του εγκλήματος γενικότερα. Ίσως και για τις ε, απάτες Κάποιος είπε ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι ίσονος σημασία. Και όμως, αν δείτε τι γίνεται στην Αγγλία, μιλάμε για εκατομμύρια λιρών. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να κάνουμε κάτι για το έγκλημα γενικότερα, συμπεριλαμβανομένε και τη απάτη. Γιατί όχι, να τα ρίξουμε όλα στο σύστημα. Και αυτά τα στοιχεία όλα μαζί να τα χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή σε έγκλημα. Χωρίς ε, πανικό για τις πολιτικές ελευθερίες. Τώρα, με την Κομισιόν Σύμφωνα απολύτω για το χρόνο τήρηση των δεδομένων. Δεν ε, θέλω να επικρίνω την εισηγήτρια, αλλά τώρα τηρούμε δεδομένα για 30 μέρες, δεδομένα τα οποία έχουμε αποκτήσει με τόσο κόπο και χρήμα, είναι νοησία. Είναι εξαιρετικό το κείμενό σα ως βάση συζήτησης, αλλά έχουμε εδώ βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ξανασυζητηθούν. Γιατί εδώ μιλάμε για το διακύβευμα, το οποίο είναι, δεν είναι άλλο παρά η ανθρώπινη ζωή. Την Κομισιόν, κυρία Βασιλιάδου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση και οι τροπολογίες πιστεύω ότι τροποποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόταση της Κομισιόν. Δεν θα εκπλαγείτε λοιπόν να σας πω ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τις περισσότερες τροπολογίες. Και ξεκινώ με το ζήτημα του περιορισμού του αντικειμένου, του σκοπού. Για την τροποκρατία όλοι είπατε ότι ναι, πρέπει να συμπεριληφθεί το σοβαρό έγκλημα. Δεν συμφωνείτε όλοι. Εγώ έχω να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση με το κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Εντάλμα Σύλληψη για ίσον σημασία έγκλημα. Εκεί η προθυμία είναι ένα χρόνο. Εδώ προτείνουμε τρία χρόνια. Τρία χρόνια, το οποίο είναι μια ουσιώδη διαφοροποίηση ω προ το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Άρα μην φοβάστε ότι πρόκειται για κλέφτε ποδηλάτων. Τώρα για το σοβαρό έγκλημα. Ορισμό. Συγγνώμη δεν άκουσα, λέει η ομιλήτρια. Σχόλιο εκτό μικροφώνου. Ορισμός ή μάλλον ο κατάλογο ορισμών του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψη είναι τα τρία χρόνια χρησιμοποιείται σε όλα τα θέματα αστυνομική και ποινική συνεργασία. Είναι κάτι το οποίο έχετε εγκρίνει και εσείς. Δηλαδή, υπάρχει στο σύστημα VIS, υπάρχει στο SIS, στο Schengen Information System. Υπάρχει στην Σουδική Πρωτοβουλία για την ανταλλαγή πληροφοριών. Παντού σε όλες τις σχετικές αποφάσεις αυτή η ρύθμιση έχει επιλεγεί γιατί θέλουμε μια συνεκτική προσέγγιση στην δικαστική και αστυνομική συνεργασία γενικότερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν νομική ασφάλεια ως προς το τι περιλαμβάνεται και τι όχι. Οι αστυνομικέ αρχές, τα κράτη-μέλη, πρέπει να γνωρίζουν με ακρίβεια σε ποιε περιπτώσει και σε ποιου τομεί μπορούν να συνεργαστούν με τι άλλε αρχέ. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εναρμονισμένη προσέγγιση στον τομέα τη δικαστική και αστυνομική εργασία. Επιπλέον, έχουμε συλλέξει όγκο στοιχείων από τα κρατημέλη αλλά και από τρίτε χώρες σχετικά με την χρησιμότητα των στοιχείων PNR τα οποία όντως συνέβαλαν στην επίλυση διαφόρων υποθέσεων. Με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, τον εισηγητή και τους, τους κοιόδης συζητήσαμε αυτόν τον όγκο πληροφοριών, κατά πόσο δηλαδή θα ήταν χρήσιμο να συμπεριλάβουμε το σοβαρό έγκλημα. Ενδεχομένως να τα ξαναπούμε με μέλη και της δικής σας Επιτροπής, μπορούμε να τα καλέσουμε να συζητήσουμε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, Η κυρία Λίχτενμπέργκερ ετοιμάζει στι τις ε, συζητήσεις, αν δεν κάνω λάθο. Οπότε θα σας ε, παρότρινα να δεχθείτε τον περιορισμό του σκοπού τη Κομισιόν. Και αυτό έχει σχέση με τι τροπολογίε του άρθρου 4 σχετικά με το πώ τύχανουν επεξεργασία στα στοιχεία, τα δεδομένα. Το άρθρο αυτό υποτίθεται αποτελεί και την ουσία τη χρήση των στοιχείων PNR. Διεπίστωσα ότι με κάποιες τροπολογίες περιορίζεται η χρησιμότητα αυτών των στοιχείων και αυτό βεβαίως θα μπορούσε να περιορίσει τα μάλλα την χρησιμότητα του μηχανισμού γενικότερα. Σας καλώ λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, να δεχτείτε την πρόταση της Κομισιόν προκειμένου. Θα περάσω ένα άλλο θέμα, το περίφημο push. Συμφωνούμε απολύτω μαζί σα, μόνο που, αυτό άλλωστε λέμε και στην πρόταση και δεν προβλέπονται εξαιρέσει. Όσον αφορά το, τα δικαιώματα των επιβατών, έχουμε συμπεριλάβει όλα τα δικαιώματα των επιβατών, των πολιτών δηλαδή, έτσι όπως τη χάνουν προστασία σε διάφορα νομικά κείμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει δικαίωμα πρόσβαση στα στοιχεία, μπορούν να ζητήσουν τη χρήση ένδικων μέσων, όλα τα δικαιώματα την χάνουν προστασίας. Προστατεύουμε και τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα όσον αφορά το ποια στοιχεία συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή το παράρτημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις υπέγραψε συμφωνία με την Αυστραλία σχετικά με την ανταλλαγή στοιχείων PNR. Ο εκεί κατάλογος είναι ακριβώς ο ίδιος. Επίσης θα υπογράψουμε σύντομα συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου ο κατάλογος, το παράδειγμα δηλαδή, θα είναι ακριβώς το ίδιο. Ο στόχος εν προκειμένου είναι με την ΙΑΤΑ και τον ΙΚΑΟ να συζητήσουμε και να εναρμονίσουμε αυτόν τον κατάλογο σε διεθνές πλέον επίπεδο. Αυτό θα έχει δύο βασικά πλέον Θα έχουμε στα χέρια μας ένα κοινό τύπο, πρότυπο μηνύματος αν θέλετε και θα είναι πολύ πιο εύκολο και πιο φθηνό για του αερομεταφορείς να στέλνουν τέτοιου είδου ειδοποιήσει. Αυτό χάρη σε μια διεθνή λοιπόν όπω είπα εναρμόνιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να διατηρήσει αυτόν τον κατάλογο στο παράρτημα, να τον εναρμονίσει και να τον κρατήσει παράλλαχτο παντού σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στι σχέσει τη με τρίτε χώρε. Διεθνώ. Όσον αφορά την περίοδο τήρηση των στοιχείων, τήρηση των δεδομένων, και εδώ εγγνώμη δίστανται. Θα ήθελα όμω να απαντήσω εν σε σχόλια τη σχετικά μου. Γνωρίζουμε βεβαίω ε, την γνωστή απόφαση στην οποία αναφερθήκατε και άλλα δικαστήρια έχουν αποφανθεί σχετικά η τήρηση των στοιχείων επικοινωνιών, ε, είναι μια πολύ διαφορετική υπόθεση σχέση με τα PNR. Δηλαδή, ο όγκο των δεδομένων των τηλεφωνημάτων μου, των γραπτών μου μηνυμάτων σε μία μέρα, οι προσβάσει μου στο ίντερνετ κλπ. Σε μία μέρα είναι μεγαλύτερος αυτός ο όγκο επαναλαμβάνω, σχέση με όλα τα PNR ολόκληρη τη ζωή μου. Υπήρχε λόγο, βλέπετε, για τον οποίο επέλεγε αυτή η λύση. Γιατί στι τηλεπικοινωνίε είχαμε πει το πολύ 6 μήνε άντε 2 χρόνια. Με τα PNR όμω τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Τα στοιχεία PNR για 6 μήνε έω και 2 χρόνια δεν μα λένε και πολλά για τι τάσει, τι τακτικέ επισκέψει ε, λαθρεμπόρων, ναρκωτικών για παράδειγμα. PNR έστω και 2 χρόνων, ακόμη και 2 χρόνων δεν σας δίνουν αρκετέ πληροφορίε. ούτε καν για την εργασία κάποιου. Λοιπόν, γιατί είπαμε πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει, ξέρετε, μαθηματικό τύπος που μας δίνει την απαιτούμενη περίοδο, αλλά είπαμε να εναρμονίσουμε τη στάση μας σε αυτό το θέμα με άλλες ρυθμίσεις που είναι για πέντε χρόνια. Έχουμε μείνει στα πέντε χρόνια γενικώ και σε άλλου τομεί δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για λόγου συνεργασία, λοιπόν, κρατάμε τα πέντε χρόνια. Θέλεις ε, να συνοψίσεις σε τρία λεπτά. Δεν θα είναι ακριβώ τρία λεπτά. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ όσο μπορώ πιο σύντομη. Αντιμετώπισα πάρα πολλά ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αύριο η ψηφοφορία, αυτό είναι σαφέ. Επομένω έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι πιστεύω ότι τα σοβαρά εγκλήματα είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν με πιο στοχευμένες προσεγγίσεις και αυτό θα είναι πιο επιτυχές. Συγγνώμη, θα τα πω στα γερμανικά να γυρίσω τον, τον ε, διακόπτη γιατί δεν ξεκίνησα καλά με τα αγγλικά. Ένα πράγμα θέλω να σας υπενθυμίσω. ως ε, αντεπιχείρημα σε αυτό το οποίο ελέγχθη. Υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη και η εμπειρία αυτή της ε, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για το τι μπορεί να κάνει κανείς με τα δεδομένα αν είναι στα χέρια μιας λάθος κυβέρνησης. Εμείς το έχουμε γνωρίσει στο πετσί μας και το ξέρουμε πολύ καλά. Γι' αυτό υπάρχει ένα κλίμα για την φύλαξη και την προστασία των δεδομένων στι ΗΠΑ που είναι πολύ διαφορετικό, διαφορετική προσέγγιση από τι ΗΠΑ ακριβώ γιατί υπάρχει η δεδομένη μα ιστορική εμπειρία. Γνωρίζουμε τι έγινε με δικτατορίες, με φασιστικά καθεστώτα, με ολοκληρωτικό καθεστώτα. Ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν, γι' αυτό έχουμε μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο σύνολο αυτό των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα σοβαρά εγκλήματα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα ορισμού, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ορισμού. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν τα ζώα θεωρήθηκαν τρομοκράτες. Αυτό τώρα μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρήθηκαν ότι οι ενέργειές τους μπορεί να έχουν τρομοκρατικό χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν είναι το δικό μου πρόβλημα εγώ θέλω να έχουμε ασφάλεια δικαίου. Δεν μας εμποδίζει κανείς <clears throat> όταν υπάρχουν αμφιβολίες και υποψίες να πάρουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια διάξηση μεταξύ μιας φυσιολογικής αρχής των διοκτικών αρχών και των μυστικών υπηρεσιών και αυτού που μπορεί να κάνει γενικά το PNR. Το PNR δεν βρίσκει τους εγκληματίες. Να μην θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυνατότητα μόνο μέσα του PNR να μάθουμε τα πάντα και να αντιμετωπίσουμε όλους τους τρομοκράτες και χωρίς αυτό δεν γίνεται. Αυτός είναι και ο λόγος <clears throat> για τον οποίο θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια αρχή για τις, ε, για τις ε, προθεσμίες θα πρέπει να εναρμονίσουμε, αλλά να εναρμονίσουμε με τη βάση της ουσίας. Τώρα, για, τους, ε, για τα σοβαρά αδικήματα, τώρα αν ένας κλέφτης ποδηλάτων είναι σοβαρό αδίκημα ή όχι, αυτό δεν νομίζω πρέπει να το συζητάμε. Εκτός της ε, τρομοκρατίας, το να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία ρύθμιση, ένα ορισμό για τα σοβαρά αδικήματα που να έχει και ασφάλεια δικαίου, Εάν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο θα ήταν θετικό, αλλά εγώ πάντα έχω υποστηρίξει την αρχή ότι πρέπει να έχουμε την ασφάλεια δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να θυμόσαστε ότι αυτά είναι δεδομένα τα οποία πηγαίνουν και αλλού. Πηγαίνουν σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλες τις χώρες τις οποίες έχουμε συμφωνίες, έχουμε κάνει συμφωνίες, αυτά τα στοιχεία πηγαίνουν και αλλού. Όπως σας είπα, εγώ θα προσπαθήσω να καταλήξω σε μια συμφωνία με αυτούς που έχουν καταθέσει τροπολογίες, να βρούμε στο βαθμό του δυνατού κάποιες τροπο, τροπολο, κοινές τροπολογίες. Στο τέλος θα καταλήξουμε σε ορισμένα θέματα, σε ψηφοφορία και θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κλείσαμε και αυτή τη συζήτηση. Ήταν πιο μακριά και από σιδηρόδρομο αυτή η συζήτηση ή από τη συζήτηση για τους σιδηροδρόμους. Και το επόμενο θέμα είναι η στρατηγική για το διάστημα. Ο κύριος Ζασάδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεισφορά τους στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές που κατέθεσαν τροπολογίες και ήρθαν σε επαφή μαζί μου για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για αυτή τη στρατηγική. Για την διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη. Λοιπόν, έχουμε το σύστημα έκνος. Γνωρίζει το Κοινοβούλιο ότι αυτή η υπηρεσία δεν είναι και τόσο χρήσιμη όσο θα έπρεπε να είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική και για τις ΜΜΕ. Το, και, και το ΕΚΝΟΣ και ο Γαλιλαίος είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συνεισέφεραν στο κεφάλαιο το σχετικό για το περιβάλλον. Μία από τις προτεραιότητες του συστήματος παρατήρησης και πλοήγησης θα πρέπει να είναι και η καταπολέμηση της ρήπανσης. Ευχαριστώ και την κυρία Φόρστερ για την συνεισφορά της, για τον τη σχέση μεταξύ αυτού του τομέα και των οικονομικών τομέων είπε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι απόλυτα δεσμευμένοι με τα διαστημικά προγράμματα και πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ και η κυρία Τικάου με τον κύριο Νταντά και την κυρία Ντουβεγάκ συνεργαστήκαμε για να μπορέσουμε να βρούμε και τη συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 1 για τη χρηματοδότηση του προγράμματος GMES. Είναι ουσιαστικό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στην έκθεση, δεν μπορούμε να το αποσιωπήσουμε. Η κυρία Δεβέρα, ο κύριος Ρίκε μου τόνισαν ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα και να έχει και τις απαραίτητες υποδομές για να το κάνει. Και αυτό να το αναφέρω στη δεύτερη συμβιβαστική τροπολογία. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ συχνά ξεχνάμε ότι η διαστημική δραστηριότητα και τα, διαστημικά σχέδια είναι πάρα πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη και για την πρόοδο των κοινωνιών μας. Ο πρώτος δικαιούχος αυτής της πολιτικής είναι ο τομέας των μεταφορών. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που εργάστηκα για αυτό το θέμα και ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν στην προετοιμασία της γνωμοδότησης. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζασάντα για το ανοιχτό του πνεύμα και για τη συνεργασία που έχει δείξει μαζί μας με τους κοιόδες συγητές εν πάση συντομία. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε τον αγνό, τον έγνος μάλλον και τον Γαλιλαίο για τα θέματα μεταφορών, για την πολιτική αεροπορία και για την υλοποίηση του συστήματος ΣΕΖΑΡ. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη απογείωση και προσγείωση στα μικρά αεροδρόμια. Το σύστημα έγνος θα πρέπει να επεκταθεί και στην, στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Ευρώπης και η πρόθεσή μου είναι να καταθέσω μια προφορική τροπολογία για να λάβουμε υπόψη τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν λειτουργεί επαρκώς καλά το σύστημα έγνος. Το σύστημα επίσης GMS θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην πολιετή χρηματοδότηση και έχω καταθέσει και μία συμβαστική τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να κατανοήσουμε και το ρόλο της διεθνούς συνεργασίας στην πολιτική του διαστήματος και θεωρώ ότι εν ώψη των πρόσφατων εξελίξεων στο διαστημικό τομέα λόγω της ρήπανσης επίσης που υπάρχει στο διάστημα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Και ένα άλλο θέμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Ζουρικέ θα πρέπει να μας απασχολήσει, συγκεκριμένα την, ε, τις μεταφορές με διαστημικά λεωφορεία που εξυπηρετούν τους διαστημικού σταθμού. Έχω καταθέσει και την τροπολογία υπαριθμών 6, μια τροπολογία μάλλον για το σημείο 6, για να έχουμε μια χωριστή ψηφοφορία, γιατί πρέπει μεν να ε, επενδύσουμε πολύ στη διαστημική πολιτική, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάμψει στο διαστημικό τομέα. Θέλουμε λοιπόν να τροποποιήσουμε και τη διατύπωση αυτής της τροπολογίας πάρα πολύ σύντομα γιατί τελειώνει, τελειώνει η συνεδρία. Τελειώνει. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μάισνερ. Θέλω ευχαριστώ. Δεν έχω καταθέσει καμία τροπολογία παρά το γεγονός ότι είμαι σκιώδη συζητήτρια. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστά αυτά τα οποία λέει ο κ. Ζασάντα. Και νομίζω ότι υπάρχουν άλλες τροπολογίες οι οποίες ε, εμπλουτίζουν το κείμενό του και θα την υποστηρίξω. Υπάρχουν άλλε τροπολογίε 5, 6, 7 και 20 οι οποίε δεν αφορούν τα θέματα μεταφορών και δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνουμε μια γνωμοδότηση η οποία επεκτείνεται σε θέματα τα οποία δεν είναι μεταφορικού χαρακτήρα. Προφανώ παίζει μεγάλο ρόλο η διαστημική στρατηγική για την ανάπτυξη σε πάρα πολλού οικονομικού τομεί και τομεί μεταφορά. Θα δούμε λοιπόν. Έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικά φιλελεύθεροι εμείς έχουμε μια ελεύθερη θέση ψηφοφορία στην τροπολογία 16 της κυρίας Λίχτεμπερκ, η οποία δεν είναι παρούσα. Προφανώς πρέπει να τεθεί μια προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της ρήπανσης στο διάστημα, αλλά δεν είναι η μόνη. Είναι πολλές οι προτεραιότητες. Εγώ λέω απλώς ότι πρέπει να αναφέρουμε όλες τις προτεραιότητες και όχι μονάχα την προτεραιότητα για την ρήπανση. Γενικά όμως, θέλω ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Ζασάδα Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε αυτή την γνωμοδότηση και είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεται το πόσο σημαντική είναι η διαστημική ε, ε, δραστηριότητα για τις μεταφορές. Φώστερο. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την συνολική συζήτηση και για την γνωμοδότηση. Από την πλευρά μας, δεν θα σχολιάσω φυσικά τα πάντα, θυμίζω ότι μας ενδιαφέρει ψηλού επίπεδου τεχνολογία, στην οποία εμπλέκονται πολλά από τα κράτη-μέλη, στις μεταφορές και αλλού φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να υποστηρίξουμε τον κλάδο. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος, τον οποίο ε, με την τροπολογία μου, σύμφωνα απολύτως ε, με το και Λέω. GMS και το ΣΕΖΑΡ. Κύριε Μάισεν, έχει δίκιο προ το εξή. Χρειάζεται κάποια ισορροπία. Ασχολούμαστε με το ΣΕΖΑΡ στην Επιτροπή μα, διότι που θα λειτουργήσει, θα μειώσει την κυκλοφορία, την ρήπανση κλπ. Χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπή προσέγγιση. Ας μην ξεχνούμε και την περιβαλλοντική πτυχή. Για τι τροπολογίε 1 και δύο, λίγο φλιαρέ, λίγο πολύπλοκε. αλλά δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Μπορώ να τι υποστηρίξω. Τώρα για την 2 τη κυρία Λίχτενμπέργκερ σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία μεταξύ του στρατιωτικού τομέα και του πολιτικού διαστήματο. Ε, δεν με νοιάζει αν κάποια κυβέρνηση θέλει να πληρώσει για όλη αυτή την τεχνολογία ε, καμία αντίρρηση, τόσο το καλύτερο θα έλεγα. Αυτό θέλουμε να βρούμε κονδύλια. Υπέρ της, μέσω της Κομισιόν ή οποιοδήποτε άλλου. Μακάρι κάποιο κράτος να μπορούσε να χρηματοδοτήσει. Τώρα, η οτιδηποτε αλλου μακαρι είναι ούτως ή άλλως πολύ σύνθετη, πολύπλοκη. Βασικά, ας βρούμε χρηματοδότηση και μετά τα άλλα λεπτομέρειες. Αυτά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ ως αντιπρόεδρος της, της ομάδας για το διάστημα. Σας ευχαριστώ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είχαμε κάνει πολύ πιο γρήγορα στο παρελθόν. Α αξιοποιήσουμε λοιπόν την υφιστάμενη υποδομή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να προχωρήσουμε, όχι μόνο για τι μεταφορέ, αλλά και για άλλου τομεί. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πολωνό συνάδελφο, γιατί το, κείμενο είναι ενδιαφέρον, είναι πυκνό, σύντομο. Στο πλαίσιο του 7ου προγράμματο πλαισίου, το οποίο συζήτησαμε, ήμουν, αν θυμάστε, εισηγητή και είχα πει ότι ο τομέα του διαστήματο και οι αερομεταφορέ είναι κρίσιμη για την επιτυχία τη Ευρώπη. Μην υπέρ λοιπόν τη τροπολογία 2 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ για την κατανομή του κόστους ε, μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα. Και τώρα όσον αφορά την τροπολογία 19, δεν νομίζω ότι ο Ανδρέας είναι σοβαρός εδώ. Βέβαια, δικαιωμά του, αλλά η προλαλήσασα ε, νομίζω το είπε. Καμία αντίρρηση. Η τεχνολογική πρόοδο σημαίνει και λιγότερη ρήπανση, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ω προς αυτό μόνοι μας. Έχουμε 10 χώρε που εκτοξεύουν δορυφόρου και διαστημικά οχήματα. Και οι άλλοι πρέπει να κάνουν κάτι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο από αυτά που μας αναλογούν. Δεν θα κάνουμε τη δουλειά για άλλους, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ και εγώ να ευχαριστώ τον κύριο Ζασάδα για την έκθεσή του και θα ήθελα να συμπεριλάβει τις τροπολογίες οι οποίες λένε ότι υπάρχει πρόβλημα σήμερα με τις διαστημικές πολιτικές λόγω του προϋπολογισμού για το 2013 χρειάζονται λεφτά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε τέτοιες πολιτικές διότι κάθε περικοπή στον προϋπολογισμό όχι μόνο σημαίνει ότι μπλοκάρει το πρόγραμμα αλλά και ότι πισωγυρίζει κιόλας Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν οι τροπολογίες που να αναγνωρίζουν το πρόβλημα και να επιμείνουν στην διατήρηση της χρηματοδότησης. Τώρα να, αυτό που λέει η κυρία Λίχτεμπεργκ ε, μας είχαν δείξει στην Τουλούζ ε, τελευταία ότι θα μπορούσαμε με την διαστημική τεχνολογία να είχαμε λύσει το πρόβλημα με το, Ιρλα... Ισλανδικό ηθέστιο το οποίο τόσα προβλήματα μας δημιουργεί. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορούμε εμείς να λύσουμε από τη γη. Γκονζάλες από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταγράφουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις για τις τροπολογίες που είναι όλες υποστηρικτικού χαρακτήρα. Ένα θέμα είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε είναι η χρηματοδότηση του GMES. Η Κομισιόν έχει κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του GMES και του Γαλιλαίου. Δεν θέλω να υπενθυμίσω τι ακριβώς λέει η Κομισιόν για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι παρακολουθείτε από κοντά αυτό το θέμα. Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι με τη διάκριση αυτή που έχει γίνει η Κομισιόν έχει τονίσει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της το κόστος του GMES μέσα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και συγχρόνως έχει στείλει ένα μήνυμα ότι θα καλύψει την ε, χρηματοδότηση του Γαλιλαίου και γι' αυτό η τροπολογία 7 μας δημιουργεί προβλήματα γιατί δίνει την εντύπωση ότι χρειάζονται οι ιδιωτικές επενδύσεις για να συμπληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει γιατί το πολιετές πρόγραμμα που έχει προτείνει η Κομισιόν θα είναι επαρκές. Μπορεί να μην καλύψει όλη την εξέλιξη των εφαρμογών, αλλά το σύστημα των δορυφόρων θα μπορέσει να συμπληρωθεί, αντίθετα από ό,τι λέει η τροπολογία σας. Ευχαριστώ κύριε Ζασάντα. Θέλετε να πείτε κάτι εν συντομία. Ευχαριστώ. Μία πρόταση μονάχα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και για τις προτάσεις σας. Χαίρομαι που έχω πάρει τόσο μεγάλη υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες και θα σας ευχαριστήσω εκ βάθους. Καρδία, σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο η ψηφοφορία, η Επιτροπή Βιομηχανίας, 22-23 Νοεμβρίου και προβλέπεται να έρθει το θέμα στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα είμαστε στο PH3 C050. Πάρτε, παρτε λοιπόν όλα τα χαρτιά σας. Είναι στο διγειτονικό κείμενο εκεί που είναι η Ολομέλεια απέναντι από την Ολομέλεια. 3C050. Η μεγάλη αίθουσα του ΕΛΚ απέναντι από την Ολομέλεια. Ευχαριστώ και στους διερμηνείς.